Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ήδη είναι 9 και τέταρτο. Πέρασε δηλαδή το ακαδημαϊκό τέταρτο που συνήθως πάντα το τηρούμε και ο κύριος Δεκάστρο επιβεβαιώνει αυτό το ακαδημαϊκό τέταρτο. Είναι ώρα όμως να ξεκινήσουμε. Είπα λοιπόν, τελείωσε και το ακαδημαϊκό τέταρτο, το επιβεβαιώνει και ο καθηγητής, ο πανεπιστημιακός, ο κύριος Δεκάστρο, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια, την εκτίμηση, την αναγνώριση και το θαυμασμό για την τόσο ταχεία υποβολή του σχεδίου έκθεσης του κυρίου Ντόρφμαν Μπράβο σας, πολύ σημαντική έκθεση και καλό παράδειγμα ότι ακολουθούμε το δρόμο του κανονισμού Omnibus. Και φυσικά παράδειγμα προς για τον ταχύ τρόπο διεκπαιρέωσης. Ε, για να επισπεύσουμε λοιπόν τη διαδικασία, ε, ο κύριος Δόρφμαν παρακάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να στείλουν στη γραμματεία ερωτήσεις με βάση τέσσερις άξονες που κατά τη γνώμη του εισηγητού είναι τα βασικά προβλήματα. Για παράδειγμα, νέα σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών μελών, περιφερειών και αγροτών ποια είναι η καλύτερη εθνική στρατηγική για την καλύτερη διακυβέρνηση ή ένα καλύτερο πρότυπο υποβολής αποτελεσμάτων για την καλύτερη διαχείριση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Πρώτος άξονας είναι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών περιφερειών και αγορατών. Δεύτερος άξονας είναι ένας έξυπνος και αποτελεσματικός τομέας ε, που θα αποφέρει καρπούς και θα προσφέρει έργο σε όλους τους πολίτες. Επίσης, πιο στοχευμένη στήριξη στον πρώτο πυλώνα. Ακόμη νιώθουμε την ε, εντύπωση της χθεσινής συζήτησης ε, από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για τον οικολογικό προσανατολισμό. Ε, επίσης έχουμε τον ενισχυμένο δεύτερο πυλώνα για ε, ζωντανές και εύρωστες αγροτικές περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, Άμεση σχετισμός με τη γεωργία. Επίσης, ε, τρίτος άξονας είναι ο θεκτικός κλάδος. Μια θεκτική γεωργία. Με πιο σταθερό περιβάλλον που ταυτόχρονα όμως θα εξασφαλίζει και την προστασία του περιβάλλοντος και θα συμβάλλει στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Πώς θα επιβραβεύσουμε τους αγρότες που μας προσφέρουν δημόσια αγαθά. Γιατί όλοι χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε αυτά τα αγαθά, αλλά δεν εκτιμούμε δεόντως την προσφορά του αγρότη. Συμβολή λοιπόν του κλάδου στην ε, και στις δράσεις για τις κλιματικές αλλαγές. Και το τέταρτο θέμα, ο τέταρτος άξονας, είναι η ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων, η διατήρηση της κοινής οργάνωσης αγοράς και η επέκτασή της ε, σε όλους τους αγρότες. Επίσης, η πρόθεση της ε, προαιρετικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Και μάλιστα ο κύριος Νταντά ασχολήθηκε εκτενώς με το θέμα αυτό. Αυτές λοιπόν οι ερωτήσεις ε, ε, διαβιβάστηκαν στους εκπροσώπους της ε, Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κύριος Μέγκελ και το επιτελείο του έδειξε μεγάλη προθυμία και διαλεκτικότητα στη συζήτηση και πολύ συνεργάσιμο πνεύμα στα πλαίσια του κανονισμού Omnibus. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στον κύριο Ντόρφμαν και κατόπιν στον Διευθυντή Μέγκελε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω, γιατί τα πιο πολλά τα είπατε. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, Προσπαθούμε να δρομολογήσουμε το σχέδιο έκθεσης για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, το οποίο και προβλέπει μέχρι το 17 Μαΐου εδώ στην Επιτροπή να έχουμε ψηφίσει. Και όντως καταφέραμε και με την ε, πολύ καλή υποστήριξη των ε, βοηθών και της γραμματείας να γράψουμε το σχέδιο της έκθεσης, το οποίο και διαβίβασα χτες ε, στους συναδέλφους ε, στην αγγλική γλώσσα. Για να δώσω στους συναδέλφους την δυνατότητα να κάτσουν να σκεφτούν ήδη και τη διατύπωση των τροπολογιών τους μετά από την παρουσίαση της έκθεσης ε, θα έχουμε σύντομο χρονικό διάστημα και προθεσμία για την κατάθεση τροπολογίων. Δεν θέλω να μπω σε θέματα ουσία στην παρούσα φάση, γιατί αυτό άλλωστε δεν αποτελεί και αντικείμενο τη σημερινή συνεδρία. Στις 12 Μαρτίου έχουμε την επίσημη παρουσίαση της έκθεση εδώ στην Επιτροπή και την πρώτη συζήτηση. Σήμερα το πρωί ουσιαστικά αυτό που είχαμε υπόψη μας ήταν να θέσουμε ερωτήσεις από πλευράς των συναδέλφων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να διαμορφωθεί με αποτελεσματικό τρόπο αυτός ο γύρος ερωταπαντήσεων είχαμε ζητήσει από τον Φράνκ να κάνει μια προετοιμασία και να ομαδοποιήσουμε κάπως αν θέλετε τις ερωτήσεις μας. Τι γίνεται, πώς είναι καταναμημένη και κατηγοροποιημένη η εκθεσή μου. Καταρχάς το νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών. Δεύτερο τμήμα της έκθεσης, ε, κλασικός πρώτος και δεύτερος πυλώνας και που εντάσσεται η διαγροτική πολιτική και ε, τρίτο θέμα, τρίτη ενότητα, ενιαίο CMO. Η κοινικό. Ε, δεν έχω λοιπόν κάτι άλλο να σας πω. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, τοποθετηθεί και στη συνέχεια να θέσουν ερωτήματα οι συνάδελφοι. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε κύριε Ντόρφμαν. Όντως μπορούμε να ζητήσουμε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Διευθυντή Μέγκελε, να μας κάνει την παρουσίαση. Νομίζω η μέθοδος που προτείνεται με την υποβολή γραπτών ερωτήσεων πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέσπευσε κατά πολύ τις εργασίες μας και τους έδωσε και πιο συγκεκριμένη μορφή και στοχευμένη. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μέγκελε ε, και αποφασίστε εσείς κύριε Μέγκελε και κάποιος άλλος από το επιτελείο σας ε, χρειάζεται να μιλήσει. Ε, <clears throat> thank you, Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντόρφμαν Έξοχη υπήρξε η συνεργασία μας μέχρι τώρα. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από πολύ στενά χρονοδιαγράμματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συγκεντρωθούμε επί των ουσιοδών ζητημάτων και πρέπει να συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για τις υποβληθείς σας ερωτήσεις. Μας βοήθησαν να προετοιμαστούμε για τη συνεδρία. Να αναφερθώ συντομία στην ανακοίνωση βάσει κάποιων διαφανειών που ετοιμάσαμε. Δεν θέλω να επαναλάβω τα υποθέντα. Θέλω να θέσω το κατάλληλο πλαίσιο. Κάνοντας το αυτό, μπορώ ήδη να απαντήσω σε κάποιες τεθήσεις ερωτήσεις των μελών. Βέβαια, θα απαντώνται και μέσω των, του, της γενικότερης ε, παρουσιάσεως. Αν έχετε απορίες, μπορείτε να βάλετε και ερωτήσεις μετά και μπορείτε να με ειδοποιήσετε αν τυχόν δεν έχω απαντήσει σωστά σε κάποιες ερωτήσεις. Δεν θα μιλήσω για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό αναλύθηκε εκτενώς από τον Επίτροπο τον κύριο Έτιγκερ χτες και είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή τη δουλειά. Η ανακοίνωση από τη φύση της ε, είναι νεολογικό κείμενο. Αναφέρεται στο πλαίσιο της πολιτικής που προετοιμάζει τις προτάσεις. Η προετοιμασία προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τι σημαίνει. Κατανομή πολιτικών αρχών της ανακοινώσεως που μετατρέπονται σε διατάξεις νομικού περιεχομένου. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κάνουν αυτό. Είναι ομαδική, συλλογική προσπάθεια. Μην περιμένετε λοιπόν να επισέλθω σε υπερβολικές λεπτομέρειες, διότι για κάποια ζητήματα Εκεί κινούμαστε ακόμα στα πλαίσια ανάλυσης και πρέπει να γίνουν και οι κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες και να ολοκληρωθούν. Θα είμαι όσο το δυνατόν σαφέστερος. Δεν αναφέρομαι στην επεξεργαστή σα πρόταση, αναφέρομαι στο κείμενο με τις ιδέες, την ανακοίνωση. Στο μέσο του θέματος βασικό στοιχείο, ένα από τα βασικά στοιχεία της ανακοινώσεως είναι η παρουσίαση ε, νέου μοντέλου ε, παράδοσης, ε, επίτευξης στόχων της κοινής ερωτικής πολιτικής. Γιατί ένα νέο μοντέλο. Διότι είδαμε ότι είχαμε εστιαστεί επί συμμορφώσεως επί σειρά ετών. Αυτό εμποδίζει τον προσανατολισμό βάση επιδόσεων και περιπλέκει την κατάσταση όσον αφορά τους θεσπιστέντες ευρωπαϊκούς κανόνες. Μια γενική προσέγγιση χωρίς μικρορυθμίσεις δεν μπορεί να καλύψει την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών με τεράστιες διαφορές όσον αφορά τις αγροτικές δομές. Έχουμε περίπλοκο νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθεί να λάβει υπόψη αυτό την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Ταυτόχρονα να πετύχει χαμηλό ποσοστό σφαλμάτων. Άρα πολλαπλασιάζονται οι κανόνες. Επεξηγήσεις, ερμηνείες, προσανατολισμοί και όλα αυτά επικρίνονται, δηλαδή περιπλέκουν την όλη εικόνα. Και αυξάνουν και το διοικητικό άχθος άλλωστε για τους συμμετέχοντες και η διέξοδος. Η αλλαγή των βασικών παραμέτρων. Δηλαδή η πολιτική να μην εδράζεται επί νομιμότητας αλλά επί επιδόσεων. Να σπάσει ο φαύλος κύκλος της ακρίβειας, της λεπτομέρειας. Ούτως ώστε να δαπανάτε σωστά και το τελευταίο ευρώ, αυτή ήταν η αρχική μέρημνα, χωρίς να βλέπουμε όμως να μην προσέχουμε κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι. Αυτό θα το αλλάξουμε. Το παλεύω, το παλεύω με τον υπολογιστή το, το νέο μοντέλο επίδειξη των στόχων. Δηλαδή, οι στόχοι της ΚΑΠ θα καθορίσουν επίπεδο ευρωπαϊκό μέσω της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τους νομοθέτες. Ο νομοθέτης θα προσφέρει στα κράτη-μέλη ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη για την υλοποίηση των πολιτικών. Στα πλαίσια βασικών απαιτήσεων, που και, αυτά, και αυτές οι απαιτήσει καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να προσθέσω κάτι άλλο και η κατανομή των πόρων. Αυτό πρέπει να γίνεται επακριβώς, με συγκεκριμένους στόχους. Να ξέρουν τα κράτη-μέλη πόσα χρήματα μπορούν να δαπανηθούν για συγκεκριμένη παρέμβαση. Σε επίπεδο 100 μελών τώρα. Ποιος είναι ο στόχος. Οι παρεμβάσεις της ΚΑΠ να ταιριάζουν στις ειδικές επιτόπιες ανάγκες. Ξεκινάμε άνωθεν και καθορίζουμε στο τοπικό επίπεδο τις ανάγκες καθορίζουμε τα στοιχεία συμμόρφωσης και επιλεξιμότητας για τους διάφορους δικαιούχους. Και έτσι κατανέμονται ευθύνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό της σφαιρικής προσέγγισης, των γενικών στόχων και των βασικών μέσων, αλλά σε επίπεδο δικαιούχων κινούνται τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το δικό τους καθήκον. Έτσι είναι απλούστερη διαδικασία, έχουν καλύτερη στόχευση τα κράτη-μέλη, καλύτερη στόχευση σε επίπεδο 100 μελών από σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αυτό στα πλαίσια στρατηγικού σχεδιασμού της ΚΑΠ βέβαια, όπου τα κράτη-μέλη αναλύουν τις ανάγκες τους, καθορίζουν στόχους και καθορίζουν τον τρόπο επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των πολιτικών επιτόπου. Εδώ έχουμε επιλόνες για το νέο μοντέλο επίτευξης των στόχων. Ξεκινάμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, Επόμενο βήμα. Ήδη παρεμβάσεω τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Συστήματα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την κυβέρνηση των δομών. Όλα αυτά ομοδοποιούνται σε ένα σχέδιο τη ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο και αργότερα γίνεται αξιολόγηση και προσμέτρηση μέσω πλαισίου επιδόσεων για να δούμε κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι διάφοροι τεθέντες στόχοι. Σημαντικό τμήμα των μέχρι τούδε συζητήσεων για την ιδέα πύρης στόχων είναι το ΚΑΠΑ της ΚΑΠ. Με την κοινή αγροτική πολιτική, έχουμε κοινή αγροτική πολιτική, θέλουμε να παραμείνει κοινή αυτή η αγροτική πολιτική. Αντίθετα με τα υποθέντα μέχρι τώρα για το σύστημα επίδειξης των στόχων, θα εξασφαλίζουμε ότι η πολιτική παραμένει κοινή βασικό στοιχείο του κοινή είναι καθορισμό στόχων Ευρωπαϊκή Ενώσεω και καθορισμό δικτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αυτό γίνεται από του νομοθέτε. Τα είδη παρεμβάσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω με βασικέ απαιτήσει, αυτά καθορίζονται από τον νομοθέτη. Οι δομέ διακυβερνήσει Ευρωπαϊκή Ενώσεω καθορίζονται και αυτέ από τον νομοθέτη. Η έγκριση τη ΚΑΠ, σχεδιασμό ΚΑΠ, εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται μια διήθηση το, που συμβαίνει σε επίπεδο 100 μελών, ούτω ώστε όλα να γίνονται στο προκαθοριστέν ευρωπαϊκό επίπεδο και πλαίσιο. Και η προσμέτρηση και η καταμέτρηση και η στάθμιση των τεκτενωμένων επιτόπου, δηλαδή κατά πώ φυσιάζουμε του στόχους, αυτό λαμβάνει η χώρα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι βλέπουμε λοιπόν. Δεν είναι ένα σύστημα που καθορίζει κάποιου στόχου, αναθέτει στα κράτη-μέλη και κάνουν τι θέλουν τα κράτη-μέλη. Το σύστημα εμπεριέχει πολλέ παραμέτρου και στοιχεία που πλαισιώνουν αυτά που πρέπει να συμβούν σε επίπεδο κράτου μέλου. Λοιπόν, το ΚΑΠΑ τη ΚΑΠ διατηρείται και προστατεύεται πολύ καλά. Τώρα στην ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει κάποιους στόχους γενικούς Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την ΚΑΠ Βλέπετε στη διαφάνεια. Πρώτα απ' όλα θέλουμε ευφύ και ανθεκτική γεωργία. Περιβαλλοντική φροντίδα, δράση για το κλίμα, συνεισφορά για την των στόχων του κλίματος και του περιβάλλοντος και θέλουμε και να πετύχουν τους στόχους για την ανάπτυξη πέθρου. Αυτοί είναι οι στόχοι που έχουν απτυχθεί περαιτέρω, μοιάζουν με τα υφετιθέντα του 2013. Στην πρώτερη μεταρρύθμιση εξελίχθηκαν περαιτέρω για ενίσχυση των πτυχών περί περιβάλλοντος και κλίματος. Και υπάρχει μια τέταρτη γενική πτυχή, στόχος, που αφορά την αύξηση της γνώσης όσον αφορά τη γεωργία. Θέλουμε περισσότερη επικουρικότητα, περισσότερη, ε, καλύτερη επίδοση και συνεργασία με άλλες πολιτικές. Και αυτή είναι άλλη μια σημαντική πτυχή στο όλο πλαίσιο. Τώρα Ανατολισμός όσον αφορά τις επιδόσεις. Οι επιδόσεις εξασφαλίζονται μέσω στόχων ευρωπαϊκών, ανέφερα τους γενικούς στόχους που καθορίζονται στην ανακοίνωση και ολοκληρώνονται στις προτάσεις με ειδικού στόχους για την ΚΑΠ, οπότε οι γενικές αρχές υποδιαιρούνται σε πιο συγκεκριμένες. Έχουμε γενικό σύνολο κοινών δικτών και αυτοί οι δείκτες είναι κρισίμου σημασία για τι απαιτήσει επιδόσεων και για τι εκθέσει και αναφορέ που πρέπει να υποβάλλουν το δεκάτη μελη Και στα πλαίσια των πολιτικών και πώ προσμετάται η απόδοση των πολιτικών. Αυτοί οι κοινοί δείκτε θα πρέπει να κατανεμηθούν περαιτέρω σε εθνικού δείκτε και στόχου που καθορίζονται σε επίπεδο σχεδίων ΚΑΠ. Είναι ο μόνος τρόπος να ελέγξουμε κατά πόσο εθνικό επίπεδο έχουν επιτευχθεί στόχοι σημαντικό στοιχείο ότι οι επιδόσεις εδράζονται στο επίπεδο κράτους μέλους και όχι σε επίπεδο δικαιούχου. Είναι σαφές ότι αν γινόταν αυτό σε επίπεδο δικαιούχου θα ήταν εξαιρετικά επαχθές. Θα επλανά το αβεβαιώτης για τον κάθε Γιώργο. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη πρέπει να συλλέγουν πληροφορίες για τις επιτόπιες εξελίξεις, να τις ομαδοποιούν να τι συμπεριλαμβάνουν σε εκθέσει που βάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε εμεί να βλέπουμε αν σε περιφερειακό εθνικό επίπεδο οι στόχοι, οι προκαθοριστέντε έχουν πράγματι επιτευχθεί. Καθήκον του κράτου μέλου ποιο είναι. Να καθορίσει το πλαίσιο για το γεωργό. Ο γεωργό να ξέρει τι πρέπει να κάνει, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει. Στα πλαίσια των διαφόρων παρεμβάσεων του σχεδίου της κοινή αγροτικής πολιτική. Βέβαια, χρειάζονται κάποιες αιρεσιμότητες προκαθοριστήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτως ώστε τα πάντα να λειτουργούν σωστά και τα κράτη-μέλη να μπορούν να εφαρμόζουν σχέδια βάσει επιδόσεων. Άλλο σημαντικό στοχείο, στο σύστημα δομών διακυβερνήσεως. Σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη στόχων σε εθνικό επίπεδο. Αυτές οι διαχειριστικές δομές, διοικητικές δομές, σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζουν τα υπάρχοντα στην ισχύουσα ΚΑΠ και όσα λειτουργούν εύρυθμα και δεν πρέπει να καταργηθούν. Και τα κράτη-μέλη δεν θα ήθελαν να γίνει κάτι τέτοιο, διότι έχουν επενδύσει πολλά στις παρούσες δομές. Αυτό σχετίζεται με την αρμόδια αρχή, που είναι κάτι σημαντικό για το δεύτερο πυλώνα και το σχετικό προγραμματισμό, την αρμόδια αρχή όσον αφορά ε, την πιστοποίηση ε, των διαφόρων φορέων πληρωμών. Άλλο στοιχείο είναι εγκεκριμένοι φορείς πληρωμών που υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη αλλά και σε κάποιες περιφέρειες και αυτοί οι φορείς κατά την κρίση μας αν θεωρούμε ότι λειτουργούν καλά δεν θα πρέπει να καταργηθούν. Είναι κρίσιμο αυτό για την υλοποίηση και για τη διαχείριση την οικονομική. Μετά, Αυτές οι διοικητικές δομές θα συμπεριλαμβάνουν κάποια συστήματα ελέγχου και διαχείρισης και πιο συγκεκριμένα το σύστημα Ajax που κατασκευάσαμε τα τελευταία 25 χρόνια μαζί με τα κράτη-μέλη και κατά την κρίση και του ελεγκτικού συνεδρίου το σύστημα αυτό λειτουργεί πολύ καλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το καταργήσουμε αυτό, διότι είναι κρισίμου σημασία για τη διαχείριση της υποστήριξης βάση περιοχών και στον πρώτο και στο δεύτερο πυλώνα. Βέβαια το Ajax, αν δείτε τους κανονισμούς, ε, υπάρχουν λεπτομέρειες αναφορές εκεί. Θα πρέπει να αφήσουμε πολλές λεπτομέρειε εκτός, που δεν θα καθορίζεται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο κρατών μελών. Επόμενο, οι φορεί πιστοποίηση που ελέγχουν τα αιτήσια λογιστικά και τι εκροέ, βασικό στοιχείο είναι η προσέγγιση ενιαίου ελέγχου, μοναδικού ελέγχου, κάτι που θεσπίστηκε προδιετία περίπου που βαίνει αυξανωμένο λειτουργικό σύστημα. δεν θέλουμε να παρατηθούμε αυτού, διότι είναι στοιχείο απλουστεύσεως, διότι σημαίνει ότι οι έλεγχοι διενεργούνται στο ενδεδειγμένο επίπεδο, αν επαναλήψεως σε άλλα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόνο χάρη, στο βαθμό των φορέων πιστοποίησεως, αν αυτοί λειτουργούν καλά, δεν θα διεξάγει τον έλεγχο σε επίπεδο εθνικό. Και αυτό θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Επίσης, στα πλαίσια των επιδόσεων. Και εδώ έχετε μια διαφάνεια που βασικά παρουσιάζει λεπτομερώς κάποια στοιχεία που βοηθούν ως αφορά την κατανόηση του συστήματος. Το διάφορο, τους διάφορους ρόλους. Τι ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι ρόλο παίζουν τα κράτη-μέλη από την άλλη. Βασικά, τι βλέπουμε εδώ. Μία σύνοψη των στοιχείων που σας εξήγησα. Μπορείτε, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά. Ξεκινάμε λοιπόν με τον ορισμό των στόχων και των δικτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Προχωράμε μετά πιο κάτω. Πάμε στο σύστημα υποβολή αναφορών, αξιολόγηση επιτεγμάτων των πολιτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και σε μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δείχνει τι θα έκαναν τα κράτη-μέλη, καθορίζουν στόχου, καθορίζουν κριτήρια επιλεξιμότητα για του δικαιούχου, ούτω καθεξής, ούτω ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πολιτική υλοποιείται επιτόπου για τους δικαιούχους. Νομίζω ότι αυτό, αυτή η εικόνα βοηθά να δει κανείς, να καταλάβει κανείς ποιοι είναι οι ρόλοι των αντιστοίχων φορέων στο όλο σύστημα. Επ' αυτής της βάσης νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αν το σύστημα υλοποιηθεί, εφαρμοστεί σωστά, θα οδηγήσει σε δομημένα σχέδια της ΚΑΠ που θα πρέπει κανονικά να είναι απλούστερα, συντομότερα και λιγότερο περιοριστικά από ότι τα παρόντα σχέδια για την κατάρτιση κανόνων. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι της συζητήσεως που διεξήχθη εδώ στην Επιτροπή αλλά και σε επαφές με τα κράτη-μέλη. Πολύ συχνά είχαν ακουστεί επικρίσεις για τα ε, πολύ μακροσκελή προγράμματα αναπτύξεως της υπαίθρου, 600 σελίδες, 800 σελίδες. Λοιπόν, διότι υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά όλα αυτά έπρεπε να υποδιαιρεθούν ε, σε λεπτομέρειες στα νέα σχέδια. Αυτή ήταν η αρχική προσέγγιση. Το νέο σύστημα ποιο είναι, ποια είναι η ιδέα. Να απομακρυνθούμε από την υπερβολική γραφειοκρατική προσέγγιση, να περιορίσουμε το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό όσον αφορά τα αναγκαία σε ένα σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από την επικουρικότητα. Τώρα να πω και κάτι για την πράσινη αρχιτεκτονική της κοινή αγροτικής πολιτικής. Εδώ πρέπει να κινηθώ κάπως αφηρημένα, διότι συνεχίζονται οι εργασίες, δεν έχουμε ολοκληρώσει το όλο σύστημα, χρειάζεται και συντονισμό μεταξύ υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας δώσω τώρα κάποια στοιχεία απλώς, μια γεύση, για να πιάσετε καλύτερα ποια θα είναι αυτή η αρχιτεκτονική. Βλέπετε την παρούσα αρχιτεκτονική. στη βάση, βασικό στοιχείο, ε, καλύπτει όλες τις εκμεταλλεύσεις, ε, είναι η πολλαπλή συμμόρφωση. Έχουμε το πρασίνισμα πάνω από αυτό και στον πρώτο πυλώνα. Ε, είναι υποχρεωτική η πολλαπλή συμμόρφωση. Το πρασίνισμα είναι υποχρεωτικό, αλλά όχι για όλες τις εκμεταλλεύσεις. Και μετά μέτρα για το κλίμα και το περιβάλλον στον πυλώνα 2, επιθελοντικής βάσης για το επίπεδο των εκμεταλλεύσεων. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία στην ανακοίνωση περί αυτού. Η παρούσα πράσινη αρχιτεκτονική θα αντικατασταθεί. Ε, το πρώτο σημαντικό στοιχείο είναι ότι πάμε σε αυτά που λέγαμε πριν για το μοντέλο για να πετύχουμε του στόχου. Εστιαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τι πρέπει να πετύχουμε. Όχι στο πώ τόσο πολύ, αλλά στο τι πρέπει να επιτευχθεί. Στόχοι για το περιβάλλον και το κλίμα που καθορίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τους στόχους τους στα πλαίσια των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ βάσει της καταστάσεως κάθε κράτους. Διότι η κατάσταση αφορά το περιβάλλον και το κλίμα ποικίλει από χώρα σε χώρα, ο κράτος μέλος, ο κράτος μέλος. Και γι' αυτό είπαμε ότι βασίζεται επί τοπικών συνθήκων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και που επιθυμεί να πετύχει ο Επίτροπος μια διαχείριση διαφόρων σχεδίων για την παραγωγή α, τροφίμων και η σωστή προσέγγιση στην Γεωργία. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε τώρα. Να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να το πετύχουμε. Και επανέρχομαι τώρα σε μια πιο συστηματική προσέγγιση. Η μελλοντική οικολογική αρχιτεκτονική θα μπορούσε να έχει αυτή τη μόρφη νέα διευρυμένη ερεσιμότητα επιτόπου. Είναι ένα στρώμα που θα μπορούσε να απλουστευτεί σε σχέση με το ισχύον σύστημα της πολλαπλής συμμόρφωσης και να συμπληρωθεί από αυτό που κάνουμε επί του παρόντος για τον οικολογικό προσανατολισμό, για το greening. Και επιπλέον θα έχουμε ουσιαστικά δύο επιλογές δεξιά έχουμε στο δεύτερο πυλώνα ε, ε, σχέδια κλιματικά και περιβαλλοντικά, αυτό που έχουμε σήμερα δηλαδή στην ΚΑΠΗ, κάτι που έχουμε αριστερά και πάλι τέτοια συστήματα ή προγράμματα κλιματικά και ε, περιβαλλοντικά στο δεύτερο πυλώνα, αλλά ένα οικολογικό τέτοιο πρόγραμμα στον πυλώνα 1. Οπότε αντικαθιστούμε το τριεπίπεδο σημερινό σύστημα από ένα διεπίπεδο με το εθελοντικό στοιχείο του πρώτου πυλώνα που θα μπορούσαν να ε, εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Αυτό το οικοσύστημα, το οικοσκήμ, το οικολογικό πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τη δυνητική αιρεσιμότητα, καταρχήν θα εξορθολογήσουμε την πολλαπλή συμμόρφωση και τον οικολογικό προσανατολισμό, τον greening, και ουσιαστικά θα τα συνδυάσουμε σε αυτό το επίπεδο της, της αιρεσιμότητας. Και μάλιστα αυτό θα γίνει με υψηλότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες από τις παρούσες και για τα δύο στοιχεία την πολλαπλή συμμόρφωση και τον οικολογικό προσανατολισμό και αυτό είναι ε, μια απέτηση ολόκληρης της κοινωνίας από την ΚΑΠ. Και θα δούμε και τα χρηματοδοτικά μέσα που θα έχει η κυνηγιορική πολιτική. Οι υποχρεωτικές, οι δεσμευτικές πρακτικές ε, σε αυτό το βασικό επίπεδο της αιρεσιμότητας θα είναι το βασικό σενάριο για πιο φιλόδοξες ε, εθελοντικές, οθελείς πρακτικές. Και εδώ επανέρχομαι σε αυτό το eco scheme, αυτό το οικολογικό πρόγραμμα που θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη δυνάμει του πρώτου πυλώνα. Η αιρεσιμότητα θα μπορούσε να παρακολουθεί τις, τη σημερινή προσέγγιση της πολλαπλής συμμόρφωσης. Δηλαδή δεν θα είναι ε, προϋπόθεση επιλεξιμότητας της ενίσχυσης, της στήριξης, αλλά μάλλον ένα σύστημα που αν ένας δικαιούχος δεν ακολουθεί τους κανόνες θα υποστεί κάποιες μειώσεις περικοπές στα κονδύλια. Και αυτό είναι κάτι σχετικά απλό και άμεσο σε σχέση με την σχετικά περίπλοκη δομή του σημερινού οικολογικού προσανατολισμού. Και μάλιστα θα ακολουθήσουμε θα επιδιώξουμε τους ίδιους στόχους ε, της πολλαπλής συμμόρφωσης, δηλαδή προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, αφήνοντας όμως μεγάλη ευελεξία στα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν τους κανόνες που θα κληθούν να τηρήσουν οι αγρότες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και θα υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών στα κράτη-μέλη για τους ε, κανόνες διαχείρισης σε σχέση με το σημερινό greening. Ακολουθώντας ε, το πνεύμα αυτού του μοντέλου προσφοράς έργου και παρουσίαση αποτελεσμάτων του delivery model που παρουσιάσαμε. Και αυτό το στοιχείο της αιρεσιμότητας θα ενσωματωθεί πλήρως στο νέο μοντέλο αποτελεσμάτων, θα συνδυαστεί και με άλλα μέσα της ΚΑΠ για το περιβάλλον και το κλίμα, γιατί το σχέδιο είναι να προβλέπει και υλοποίηση και περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, οπότε ο τρόπος που θα διαμορφώσουμε την αιρεσιμότητα θα εξαρτηθεί και από τις φιλοδοξίες μας και τους τρόπους που θα προγραμματίσουμε τις ενισχύσεις του δεύτερου πυλώνα. φυσικά θα, θα συνδυαστεί με αποτελέσματα και ποσοτικοποιημένους στόχους, θα ανήκει στο σχέδιο της, της ΚΑΠ και θα συνδυαστεί με αποτελέσματα και ποσοτικοποιημένα αποτελέσματα ε, εν ώψη και των πολιετών προοπτικών. Πολλές ε, ερωτήσεις ε, αναφέρθηκαν για τα μέσα της κοινής οργάνωσης αγοράς, όπως είπε ο κύριος Ντόρφμαν. Γι' αυτό το ζήτημα υπευλέθησαν πολλές ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά τις δικλείδες ασφαλείας, τα δίκτυα ασφαλείας που είναι τα μέτρα παρέμβασης όπως δημόσια και ιδιωτική αποθεματοποίηση, ε, τα μέτρα για την κρίση και τα έκτακτα μέτρα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι λόγω της φύσης τους δεν μπορούν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων. Είναι μηχανισμοί και μέσα που χρησιμοποιούνται δυνάμει της κατάστασης που παρουσιάζει η αγορά. Οπότε μια διαρθρωμένη διαδικασία προγραμματισμού που θα οδηγήσει σε ένα σχέδιο της ΚΑΠ δεν προσαρμόζεται σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις στην αγορά. Οπότε δεν μπορεί να εμπίπτει στο delivery model και το σχέδιο της ΚΑΠ. Το ίδιο ισχύει και για τα αμυγός κανονιστικά σκέλη της, ε, του κανονισμού ΚΟΑ, όπως προδιαγραφές ε, θέσεις εμπορία. Αυτό δεν έχει σχέση με τη δαπάνη ε, ή τις δραστηριότητες στήριξης. Αφορά την κανονιστική πολιτική και θα πρέπει να παραμείνει και που είναι, να μην ενταχθεί δηλαδή στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Και νομίζω ότι έτσι διασκεδάζουμε και κάποιες ανησυχίες που διατυπώθηκαν και που είπαν ότι αν τα αφήσουμε όλα στα χέρια των κρατών μελών θα υποβαθμιστούν οι κανόνες περί ή κάποιες προδιαγραφές. Αυτό δεν ισχύει, γιατί αυτό θα παραμείνει στο επίπεδο το σημερινό. Δεν θα μεταφερθεί στο σχεδιασμό. Άλλα είδη όμως παρέμβασης αγορά που σήμερα καλύπτονται από την κοινή οργάνωση αγορά, ίσω περιληφθούν στο delivery model και στο, στη διαδικασία σχεδιασμού. Και αυτά κάνουν ουσιαστικά οι οργανώσεις ε, παραγωγών. Τα επιχειρησιακά προγράμματα ακριβώς ακολουθούν την ιδέα της επικουρικότητας. Όπως ε, φαίνεται και στο μοντέλο περί αποτελεσμάτων, περί παρουσίασης έργου, του delivery model. Θα μπορούσαν τώρα να μεταφερθούν στην διαδικασία προγραμματισμού σε συνδυασμό με άλλα μέσα στήριξης που σας παρουσίασα προηγουμένως και θα στηρίζονται σε γενικούς και ειδικούς στόχους στο σχεδιασμό και στο στόχους του σχεδιασμού της ΚΑΠ και σε δείκτες και στόχους παραγωγής. Επί του παρόντος δεν μπορώ να πω και τίποτα παραπάνω για τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση αγοράς και την αλληλεπίδραση του με το νέο μοντέλο παρουσίαση αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης του delivery model. Τώρα, τα τελευταία μου σχόλια θα περισταθούν γύρω από δύο θέματα που καλύπτονται στις ερωτήσεις. Καταρχήν, η σχέση αυτού του εχειρήματο με την πιθανή πρόταση που θα, κάνει, θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα UTP στις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018 αναφέρεται αυτή η πρόθεση ε, και κανονικά αναμένεται ως ξεχωριστή πρόταση για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και όχι ως τμήμα των προτάσεων για την ΚΑΠ μετά το 2020. Και αυτό γίνεται γιατί θεωρούμε ότι η πρόταση για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές μπορεί να δρομολογηθεί και να διεκπαιρεωθεί πριν τα τέλη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Και άρα οι νέοι κανόνες για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές να τεθούν σε εφαρμογή νωρίτερα. Ενώ οι κανόνες για την ΚΑΠ μετά το 2020 θα τεθούν σε ισχύ μετά το 2020. Είναι αυτονόητο. Δεν έχει νόημα λοιπόν τις αθέμετες εμπορικές πρακτικές να τις εντάξουμε σε ένα ευρύτερο πακέτο που θα τεθεί σε εφαρμογή πολύ αργότερα ενώ έχουμε τη δυνατότητα να τις εφαρμόσουμε πιο γρήγορα. Στα πλαίσια της εσωτερικής μας ε, προσπάθειας να βελτιώσουμε την θέση των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων αφορά το θέμα της διαφάνειας, ε, διαφάνειας και προσδιορισμού των τιμών. Και εδώ ε, ξεκινούμε από την ιδέα ότι οι βασικοί κανόνες που θα, εφαρμόζονται θα μπορούσαν να δορυπηθούν με βάση κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Δεν χρειάζεται να αλλάξει ο βασικός κανονισμός ή οι βασικοί κανονισμοί. Και όταν υποβάλουμε τις προτάσεις αυτές σε κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις θα μπορούν να τεθούν σε ισχύ σχετικά γρήγορα. Δεν χρειάζεται και πάλι να περιμένουμε το ευρύτερο πακέτο που θα τεθεί σε ισχύ μετά το 2020, δηλαδή το 2021 και μετά. Αυτά κύριε Πρόεδρε Αυτά είχα να σας προσφέρω σήμερα ως γενικές πληροφορίες. Ελπίζω να κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις και απορίες σας και αν δεν τα κατάφερα έχουμε και τώρα το χρόνο να επανέλθουμε σε επιμέρους ζητήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μέγκελε. Αυτή είναι μια νέα ποιότητα α, της προσπάθειας. Ότι για μερικές α, πράξεις που είναι πιο απόμακρες αφορούν πιο απότερο ε, μέλλον. Έχουμε και την φάση για τις, τις των εφαρμοστικών και κατεξουδότηση ε, πράξεων, που είναι πιο άμεσης εφαρμογής. Επίσης ε, είχαμε και συνεργασία, είχατε και συνεργασία με τα κράτη-μέλη και όχι μόνο σε επίπεδο Υπουργείων, αλλά και σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους. Αυτά και περάμε στη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, και ο εισηγητές για τρία λεπτά και στους υπόλοιπους για δύο λεπτά. Έχουμε αρκετό χρόνο, όχι απεριόριστο βέβαια, αλλά επειδή είναι σημαντικό το θέμα, καλό θα είναι να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για τις ομιλίες. Η κυρία Αγγιλέρα πρώτα. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχήν θέρμα τον κύριο Ντόρφμαν γιατί πραγματικά τήρησε την υπόσχεσή του να υποβάλει όσον όπο την ε, έκθεσή του και με την ταχύτητα αυτή μας διευκολύνεται και εμάς ε, και με την προθεσμία για τις τροπολογίες. Χαιρετίζω λοιπόν την προσπάθειά του και την τήρηση της υπόσχεσης που έκανε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει γρήγορα το σχέδιο έκθεσής του. Η Ισπανία, η πατρίδα μου, θα εξετάσει αυτό το μοντέλο νέας σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Και εκεί που υπάρχουν ε, ε, σαφείς ρυθμίσεις του συντάγματος, ώστε στα, και στα γεωργικά ζητήματα στη χώρα μου να έχουμε και άλλα επίπεδα. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά σχέδια, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι όντως εθνικά, αλλά ίσως κάτι τέτοιο έχει έρθει σε αντίφαση με την συνταγματική εθνική τάξη... για την κατανομή, κατομερισμό των αρμοδιοτήτων. Ίσως λοιπόν αυτό δημιουργήσει κάποια πρόβλημα σε κάποια κράτη-μέλη. Γιατί έχουμε τα σχέδια, αλλά δεν μπορούμε για όλα τα επιμέρους σημεία να έχουμε εθνικό μόνο σχεδιασμό σε περίπτωση που η ένωμη τάξη προβλέπει διαφορετικό κατομερισμό αρμοδιοτήτων. Ε, η επιλογή των νέων αποδεκτών της ενίσχυσης, των νέων δικαιούχων της ενίσχυσης του πρώτου πυλώνα θα παραμείνει με βάση τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μείνει αυτός ο προσδιορισμός των δικαιούχων στα χέρια των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, ε, στα κράτη-μέλη θα αρχίσει να διαμορφώνεται περισσότερο η έννοια του ενεργού αγρότη ανάλογα με την αγροτική δραστηριότητα που θα έχει ε, τη διατήρηση όχι των ιστορικών δικαιωμάτων. Πάντως, αν ο ορισμός του συγκεκριμένου δικαιούχου, του συγκεκριμένου αποδέκτη, θα συγκεκριμενοποιείται σε επίπεδο κρατών μελών, αυτός ο προσδιορισμός, αυτή η αναγνώριση του αποδέκτη, ίσως και πάλι δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί μπορεί να ορίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους στόχους, αλλά ε, ο συγκεκριμένος προσδιορισμός σε επίπεδο κρατών μελών ίσως δημιουργήσει κάποια στρέβλωση. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι οι παρόντες δείκτες αποτελεσμάτων είναι ξεπερασμένοι, τουλάχιστον κατά 5%. Και έχουμε μια μεταρρύθμιση που θα δράζεται περισσότερο στα αποτελέσματα. Οπότε τι θα γίνει, θα έχουμε νέου νέους αποτελεσμάτων. Φαντάζομαι ναι, αφού οι παλιοί είναι παροχημένοι. Και είπατε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την γραφειοκρατία, να πλουστεύσουμε την κατάσταση και παρόλα αυτά θα έχουμε τελείω νέου δείκτε αποτελεσμάτων. Επίσης, αυτή, αυτή η νέα κατανομή για τα περιβαλλοντικά θέματα φαίνεται καλύτερη, γιατί όλοι επικρίνουμε το greening, αλλά εδώ έχω κάποιες αμφιβολίες. Θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικές ε, αγορές μεταξύ των κρατών μελών έχοντας διαφορές στις περιβαλλοντικές τους φιλοδοξίες. Γιατί πώς θα χρησιμοποιηθούν οι ΚΟΑ. Θα μπορούσαμε εκτός από οικονομική ανταγωνιστικότητα να έχουμε και περιβαλλοντικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σένορα, Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας τον κύριο Ντόρφαμ που ήδη μας υπέβαλε το σχέδιο έκθεσής του. αφού μας το ζήτησε, ούτε και εγώ θα επισέλθω σε λεπτομέρειες της πρότασης. Θα επικεντρωθώ μόνο στις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε και πάλι την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχε και πάλι την αίσθηση ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια προσβολή στην νοημοσύνη μας. Ακούγεται υπερβολικό αυτό που λέω και απότομο, αλλά συνεχίζουμε τις συζητήσεις και τα λόγια χωρίς να έχουμε καμία συγκεκριμένη πρόταση για να δώσουμε μια απτή λύση στο ουσιαστικό πρόβλημα που έχουμε. Και το ουσιαστικό πρόβλημα που έχουμε είναι η ίδια επιβίωση χιλιάδων ε, ε, ε, οικογενειών γεωργών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή ενισχύει την επισφαλή θέση των αγροτών και των αγροτησών και επιτρέπει την επέλαση μιας ρηπογόνου βιομηχανικής πολιτικής στη γεωργία, μιας εντατικής δηλαδή γεωργίας ενώ υποτίθεται ότι ε, η γεωργία θα βοηθήσει την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντρυφήσει και να εξετάσει ενδελεχώς τις επιπτώσεις της ΚΑΠ. Γιατί είπαμε ότι θέλουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα των χαμηλών γεωργικών εισοδημάτων, ε, αλλά αυτό δεν το συνδέουμε με τις ε, επιπτώσεις της μέχρι τώρα κοινής γεωργικής πολιτικής. Ποιος είναι ο υπέτειος για τη σημερινή κατάσταση. Θα πρέπει να μας το εξηγήσετε. Ποιος είναι ο υπεύθυνο. Γιατί αν είναι άσχετη η ΚΑΠ με τη σημερινή κατάσταση, τότε ποιος έκανε τη διαχείριση. Ποια πολιτική ε, μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Ποιος ε, επινόησε την πολιτική που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση. Έχω και άλλη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την υπερπαραγωγή, τα πλεονάσματα και τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες αντιλήσατε κάποιο δίδαγμα από τελευταίο εμβληματικό μέτρο που ήταν η οικειοθελής μείωση της γαλακτοκομικής παραγωγής, όταν τη σήμερα ημέρα στο, στις συζητήσεις ε, με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών αγνωρίσατε την ε, μεγάλη υπερπαραγωγή γάλακτος που έχουμε σε πολλά και τα πολλά πλεονάσματα. Τι αποτελεσματικότητα είχαν αυτά τα δημόσια κονδύλια με τα οποία προσπαθήσατε να μας πείσετε ότι θα δώσουν τη μαγική λύση για την ε, κατά της υπερπαραγωγής. Πού είναι η αποτελεσματικότητα. Δεν είναι καλύτερα να μιλήσουμε για ρύθμιση, για παρέμβαση στην αγορά. Δεν είναι καλύτερο να βελτιώσουμε τις τιμές παραγωγού και αυτό το θέμα να το βάλουμε στο επίκεντρο της ΚΑΠ. Δεν θα ήταν καλύτερο να μιλήσουμε για ένα γεωργικό μοντέλο που δεν θα ρηπαίνει το περιβάλλον, αλλά θα παράγει υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα. Δεν είναι καλύτερο να εστιάσουμε σε αυτά τα σημεία τη συζήτηση και να σταματήσουμε αυτή την απάτη, να σταματήσουμε να ξαπατούμε και να ξεγελάμε την κοινωνία με μια κοινή γεωργική πολιτική που σε τελική ανάλυση το μόνο που κάνει είναι να συγκεντρώνει τα δημόσια κονδύλια και το πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια. Δεν πιστεύετε ότι μια ουσιαστική αλλαγή θα ήταν η λύση και για τους αγρότες και για, τις, ε, για την κοινωνία. Σταματήστε να μας κοροϊδεύετε. Έχουμε βαρεθεί. Έχω επιβδίσει. Από το 1994 χρησιμοποιείτε όλα αυτά που θέλει ε, να αλλάξει η κοινωνία για να συγκαλύψετε κάποιες, ε, προτε... κάποιες πρωτοβουλίες που ουσιαστικά το αντίθετο αποτέλεσμα επιδιώκουν. Σταματήστε πια να μας κοροϊδεύετε και να μας ξεγελάτε. Ευχαριστώ. Κυρία Σέρα, σχεδόν συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, με εξαίρεση αυτό που είπα ότι θέλουμε να ξεγελάσουμε τους αγρότες. Δεν ξέρω η Επιτροπή εμείς, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε ή να ξεγελάσουμε τους αγρότες. Αλλήμωνο, εμείς το αντίθετο, θέλουμε να εξυπηρετήσουμε, να βοηθήσουμε τους αγρότες. Αλλά ως προς το πρώτο σκέλος ε, της ομιλίας σας, θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει να βρούμε λύση και για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να φέρουμε τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, στο επίκεντρο και να δούμε πώς μπορούμε να τις συνδέσουμε με το greening και πώς μπορούμε να εντάξουμε και τις μικρές εκμεταλλεύσεις ε, σε αυτή τη διαδικασία του οικολογικού ε, προσανατολισμού. Γιατί δεν είναι χιλιάδες αυτές οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είναι εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολλές. Μεγάλη πρόκληση αυτή σημαντική. Κυρία, ο κύριος μάλλον Βάιτς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολλά κύριε Ντόρφμαν για την ε, βάσει αυτή των εργασιών μας ε, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ίσως ε, αμελήσατε την άμεση θέση στην αμπορία ως στόχο σε ό,τι αφορά την ε, αλυσίδα παραγωγής και σε ό,τι αφορά τους μεγάλους παραγωγούς στην, παράδο, στην παράγραφο 18 να πω ότι δεν μπορούμε να έχουμε μόνο ένα ελάχιστο πόσο για την οικολογική προσέγγιση των εκτάσεων. Θα πρέπει να δούμε και τα μέγιστα ποσά προς την κατεύθυνση αυτή. Και μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει το άρθρο 25, όπου μιλάτε για την, ε, τις και τι δυνατότητε της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Να κάνω μια ερώτηση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πιστεύετε ότι η χρήση ευρωπαϊκών πόρων, των πόρων των φορολογούμενων ουσιαστικά θα πρέπει καταρχάς να ωφελεί τους Ευρωπαίους γεωργούς και καταναλωτές και δεν είναι η δική μας ε, αρμοδιότητα να κοιτάξουμε τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Γεωργία, αλλά βασικά να προστατεύσουμε από την παγκοσμιοποίηση τους Ευρωπαίους ε, γεωργούς ε, για την επαναθνικοποίηση τώρα, όπως ονομάζεται. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ασφάλως το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, χαίρεται που διαρκώς κατηγορείται για τη γραφειοκρατία, για την έντονη γραφειοκρατική διαμόρφωση της όλης της διαδικασίας και καταλαβαίνω προφανώς ότι καλό θα ήταν αυτές οι, θα ήθελε μάλλον αυτές οι διαδικασίες να α, ρυθμίσονται σε επίπεδο 28 κρατών μελών. Το κατά πόσον όμως οι 28 καινούργιε γραφειοκρατίες θα είχαν αποτέλεσμα λιγότερη συνολική γραφειοκρατία συνολικά για όλη την Ευρώπη, αυτό πραγματικά το, με, με, το αμφιβάλλω. Και σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, καταλαβαίνω ποιε είναι οι συνέπειε. Αυτό τι σημαίνει όμω για μικρομεσαίε χώρε, ε, όπου για παράδειγμα έχουμε τέσσερι ε, χώρε, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία κτλ. Τι σημαίνει ο, αν οι γεωργοί έχουν διαφορετικά συστήματα ενίσχυσης σε τόσο στενή γεωγραφική απόσταση, όπου ουσιαστικά είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός. Πώς ε, θα εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει σωστός ανταγωνισμός και όχι στρεβλός. Εγώ έχω μεγάλες αμφιβολίες ε, αν ε, στη μία χώρα οι ενισχύσει είναι ύψου εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και στην άλλη χώρα, λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, οι ενισχύσει είναι σε ύψο εκατομμυρίων. Πραγματικά πολύ αμφιβάλλω. Θα ήθελα να τοποθετηθείτε από αυτού. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τους και ηγητές και περνάμε στους υπόλοιπους βουλευτές για δύο λεπτά οι εκτός από την κυρία Ντελαγέ που θα έχει απεριόριστο χρόνο ομιλίας. Και θα έχει απεριόριστο χρόνο ομιλίας η κυρία Ντελαγέ γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Και της ευχόμαστε χρόνια πολλά και το δώρο μας είναι μπορεί να μιλήσει όσο θέλει, ενώ οι υπόλοιποι μόνο δύο λεπτά. Παρακαλώ κυρία Ντελαγέ. Και χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ, θα καταχραστώ του χρόνου, Πρόεδρε. Καταρχάς αφορά την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε μελέτη αντικτύπου όσον αφορά το μηχανισμό New Delivery και εκπίσω από τη μέθοδο. Βλέπω κάποιου κίνδυνου. Ο πρώτο είναι ο εξή. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει επικουρικότητα δεν ισότητα με επανεθνικοποίηση, εγώ όταν πέραμε θεωρία στην πράξη, Δυστυχώ δεν είμαι τόσο πεπισμένη. Μια άλλη ανησυχία, κίνδυνο για μένα, είναι η απόσταση των εξουσιών του συνομοθέτη που είμαστε εμείς μέσω του εγχειρήματο που κάνουμε για την ΚΟΑ και δεν βλέπω στην πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η κατεξοδότηση πράξης. Δηλαδή, εμεί μόνο βασικέ αρχέ μπορούμε να καθορίσουμε και σταματάμε εκεί. Σαν συνομοθέτη, ενοχλούμε από αυτό. Άλλο κίνδυνο, τρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών σε εθνικό, στα εθνικά σχέδια. Το βλέπουμε αυτό μέσω το θέματο τη περιφερειοποίηση. Αλλά φοβάμαι μήπω αυτό η προσέγγιση ενισχυθεί ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Μια ΚΑΠ πιο απλουστευμένη, τον ριβόμαστε όλοι. Δεν είμαι σίγουρος εάν τελικά αυτή την πρόταση την ελοπίσουμε ε, ότι θα πετύχει αυτό μετά το χρονοδιάγραμμα να, να περάσουμε στη μεταρρύθμιση ε, αυτή μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογέ μου φαίνεται ότι δεν είναι πολύ λογικό για το Omnibus που ήταν απλώς ένα εγχείρημα που αφορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειαστήκαμε 13 μήνες. Η τελευταία μεταρρύθμιση δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα σε όλα τα κάτι μέλη. Πολλοί γεωργοί διαδηλώνουν σήμερα στην ε, Γαλλία εδώ και 15 χρόνια για τον χάρτη των διαφόρων περιοχών των γεωργικών που βρίσκονται σε μενικτική θέση και τώρα να του πούμε ότι θα κάνουμε και άλλη μεταρρύθμιση. Έχουν κουραστεί από αυτή τη συνεχή αλλαγή. Δώστε μα το χρόνο να κάνουμε μια πραγματική μεταρρύθμιση. Η οποία μεταρρύθμιση θα είναι χρονικά πιο σταθερή. Τελευταίο σχόλιο όσον αφορά την ίδια την έκθεση του συναδέλφου Ντόρφμαν. Είναι καλή έκθεση. Πολλά σημεία που ανέφερα συμπεριλήφθησαν σε διάφορου παραγράφου εκθέσεώ του. Δεν υπάρχει παρά μόνο ένα πρόβλημα για μένα που ισχύει και για την ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που θα πω η λέξη επένδυση δεν εμφανίζεται πουθενά. Αυτό με λυπεί. Εάν έχουμε φιλοδοξίες για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, πιστεύω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε όσον αφορά την επίτευξη αυτών των φιλοδοξιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα πω κάτι και να με συμπαθάτε, αλλά οι, διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες των αγρότων ε, έχουν κάποιο νόημα για αυτούς που χαράζουν τις πολιτικές, γιατί τους επισημαίνουν τα προβλήματα. Ο κύριο Σέγγε, ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντόρφμαν για το σχέδιο της έκθεσης το οποίο το διάβασα με πολύ ενδιαφέρον χθε το βράδυ. Κάποιες παρατηρήσεις επιτρέψτε μου. Η ΚΑΠ ε, επί δεκαετίε. Ε, καθόρισε τις τιμές των τροφίμων και όθησε τις μεγάλες επιχειρήσεις στο καλό δρόμο, αλλά τι τίμημα πληρώσαμε. Η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική οδήγησε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε οικονομικό θάνατο. Οι μεγάλες άμεσες ενισχύσεις οδήγησαν σε απώλεια βιοπικιλότητας, μονοκαλλιέργειες, μεγάλες απώλειες και τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν σταθερά για σκάνδαλα σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ζητήματα μικροβιακής εντοχής, να μην ξεκινήσω καν να μιλάω. Οι πολίτες λοιπόν της Ευρώπης ε, θέλουν πιο πολύ ποιότητα στα τρόφιμα. Και οικολογικό και κοινωνικό προσανατολισμό και μάλιστα με προσμετρήσιμες επιδόσεις. Μία πολιτική η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους ε, γεωργούς ε, να αντιμετωπίσουν τους φυσικούς πόρους με υπεύθυνο τρόπο, να εφαρμόζουν τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους χωρίς να ε, πάσχουν οικονομικά σε ό,τι αφορά το εισόδημα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σωστοί κανόνες και σωστά οικονομικά κίνητρα με τη διάθεση των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πόρων. Κύριε Ντόρφμαν, λοιπόν, έχετε την τόλμη και το θάρρος για ένα πιο φιλόδοξο κείμενο, το οποίο θα πει τα πράγματα με το όνομά τους, τα προβλήματα με το όνομά τους, γιατί λίγο πολύ θεωρώ ότι η πρότασή σας ε, κινείται στο status quo και μια κουβέντα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ε, εκτενή αυτή παρουσίαση σε ό,τι αφορά την τις προτεραιότητες. Αναφέρεται προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος, αλλά για την ευημερία των ζώων, την προστασία των ζώων δεν άκουσα τίποτα. Δεν ε, τρέπεστε. Γιατί το βαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχετική μελέτη που έδωσε εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ε, κατάδειξε ότι 80% των πολιτών θέλουν πιο πολύ προστασία των ζώων. Και εσείς τι κάνετε, μας αφήνετε στο κοινό για μια φορά ακόμη. Δεν είναι τρόπος, πιστεύω, αντιμετώπισης ε, της βούλησης των πολιτών εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όταν εξαντλείτε το δίλεπτο, ρίχνετε και μια ματιά προς τον πρόεδρο και το εργαλείο του, που είναι το σφυράκι του Ρίχνετε και καμιά ματιά προς τον Πρόεδρο. Ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Ντόρφμαν, ο συνάδελφός μας, έχει κάνει εξαιρετική, τέλεια δουλειά. Τώρα, το δικό μας καθήκον είναι να το βελτιώσουμε και να το ολοκληρώσουμε, να το ριστικοποιήσουμε το έργο του αυτό. Χθες, εδώ, στην αίθουσα, στην Επιτροπή μας, συζητήσαμε για την ανάγκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υπάρχουν δεύτερης κατηγορίας ε, πολίτες. Την προηγούμενη ημέρα παρουσίασα μία αναφορά και ένα αίτημα της ε, Λιθουανικής ε, Γεωργικής Ένωσης για να μην υπάρχουν πραγματικά πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι γεωργικές πληρωμές για το 2021 για τους αγρότες να μην είναι πιο χαμηλές από το μέσο όρο του 2010, ενώ οι ενισχύσεις για την πράσινη προσέγγιση θα πρέπει επίσης να συνεχιστούν. Νομίζω ότι το έγγραφο λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το θέμα αυτό απασχολεί ιδιαίτερο τους πολίτες και τους αγρότες μας. Για την επόμενη περίοδο λοιπόν θα πρέπει να το επιλύσουμε το θέμα αυτό και όχι να συνεχίσουμε επαόριστον τις συζητήσεις. Αν οι αγρότες δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν, Πώ θα διαμορφωθεί ο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι, θεωρώ, φυσιολογικό να εξαναγκάζονται οι αγρότες να πάνε σε άλλες χώρες για να εργαστούν στον αγροτικό κλάδο. Αυτό θα πρέπει, θα πρέπει να τραυματιστεί ω πρακτική. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιβίωση στη χώρα του καθενό. Και όπω είπαν και οι συνάδελφοι, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πολιτική θα πρέπει να παραμείνει ενιαία, μία και μοναδική. Όχι 27 κατακρεματισμένα κομμάτια, όπως προσπαθεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποποιηθεί των ευθυνών τη και να θέσει όρους για τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι είναι πολύ διαφορετικέ οι συνθήκε που επικρατούν στα κράτη-μέλη και αν ακολουθήσουμε την τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Όντω, έχετε δίκιο ότι τα προβλήματα πρέπει να τα επιλύουμε και όχι μόνο να τα διαπιστώνουμε. Ο κύριος Χόισλινγκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντόρφμα για την παρουσίασή σας, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να απαλλαγώ από την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα καταφέρνει και τα κρατή και η ευγεωργική πολιτική ε, είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας και θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν. Νομίζω ότι παρουσιάσαμε όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Δεν αμφιβάλλουμε. Δεν αμφιβάλλουμε ότι θέλουμε να περάσουν όσο δεν πέρασαν στην προηγούμενη γεωργική πολιτική. Γιατί όμω τι περιμένετε πραγματικά να τα εφαρμόσουν αυτά τα κράτη-μέλη. Χτε αναφέρθηκαν δύο στοιχεία στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου και την παρουσίαση του κ. Oettinger. Εσείς κάνετε Λες και δεν τα ακούσαμε όλα αυτά και είπατε ότι 80% των ε, εκτάσεων θα υπαχθούν στην διαδικασία της πράσινης προσέγγισης. Χθες όμως ακούσαμε ότι είναι 5 αυτό το ποσοστό. Θεωρώ ότι τα βλέπετε τα πράγματα αεροποιημένα. Και τώρα θέλετε να γίνει αυτό σε επίπεδο κρατου μέλους. Εγώ πολύ φοβάμαι και όχι μόνο εγώ, ότι ο ανταγωνισμό σπρώχνει τις συνθήκε ε, προ τα κάτω, δηλαδή επικρατεί ο λιγότερο φιλόδοξο και όλοι φοβούνται από πλευρά των κράτων μελών ότι θα έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα οι αγρότε τους αν θέσουν πιο υψηλου όρου, Μα πώς θα περάσουν τότε φιλόδοξοι ε, περιβαλλοντικοί στόχοι και αυτό το ερώτημα δεν το έχετε απαντήσει ακόμα. Ωραία, μία χώρα θα ένα στόχο, τον ελέγχει τον στόχο μετά από κάποια χρόνια, διαπιστώνει ότι έχει πετύχει ή δεν έχει πετύχει μάλλον το στόχο. Και τι θα κάνει στην περίπτωση αυτή, θα επιτρέψει τα χρήματα, θα τα παρέπω από τους αγρότες, όπως και σε όλες τις άλλες περιβαλλοντικές μεταγραφές που θέτουμε στην Ευρώπη. Στη τελική ανάλυση τι λέμε, Ωραία, δεν πετύχαμε το στόχο μα. Τι κάνουμε, δίνουμε μια παράταση στην προθεσμία και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Μια τρύπα στο νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απλά στο εκεί και παρατείνει τις προθεσμίες χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένες συνέπειες. Το τελευταίο θέμα με μπέρδεψε. Είπατε πράσινο, πρασινίσμα στον πρώτο πυλώνα με πολλαπλή συμμόρφωση, αλλά όχι για όλους. Και τα περιβαλλοντικά μέτρα μόνο στο δεύτερο πυλώνα. Μετά είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, συγκεκριμένη διατύπωση των στόχων ε, ως προτεραιότητα. Και ότι τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν αυτό. Όλα αυτά μου προκαλούν μια κάποια σύγχυση. Γελάτε, καταλαβαίνω. Αλλά ο Επίτροπος στην τελευταία συναντρίαση γελώντα, μα είπε ότι εντάξει, περιμένετε λίγο να αντευκρινιστεί η κατάσταση. Αν θέλετε να τα πετύχουμε αυτά σε μισό έτος, σε μισό χρόνο, θέλουμε πιο συγκεκριμένε απαντήσει όχι γυναικολογίες. Τρία λεπτά μιλήσατε κύριε Χόισλινγκ. Ε, μάλλον θα καλέσω τον κύριο Μέγκελ να κάτσει δίπλα μου για να ρίχνετε και καμιά ματιά προς το Προεδρείο. Γιατί όλοι κοιτάτε τον κύριο Μέγκελ και κανένα τον Πρόεδρο και το σφυράκι του. Ο κύριος Κάστρο, καταρχάς έξοχη δουλειά αυτή του συναδέλφου Ντόρφμαν. Διάβασα την έκθεση και επί πολλών σημείων ε, συμφωνώ. Εγώ θα ενίσχυα το κομμάτι που ο συνάδελφος υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί, να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση. Ε, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Μάρτιν Όσλιμ, ε, δηλαδή χρειάζεται μια μεγάλη διαδικασία απλούστευσης. Αλλά η απλούστευση αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα κράτη-μέλη οι περιπλοκές δεν θα αυξηθούν, θα πολλαπλασιαστούν. Και όπως έλεγε η Κλάρα Αγγιλέρα, σε χώρες που έχουν μία οργάνωση περιφερειακή, πώς θα καταφέρουν να χειριστούν ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, διότι κατά κάποιο τρόπο είναι σαφές από την ε, παρουσίαση του Διευθυντού κ. Μέγκελ ότι συμπεριλαμβάνεται το σχέδιο ανάπτυξη πέθρου για την ανάπτυξη πέθρου οι χώρες που έχουν μια οργάνωση περιφερειακή δεν θα το βρουν εύκολο να φέρουν σε εθνικό επίπεδο αυτό που ήδη σήμερα είναι σε περιφερειακό επίπεδο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος στην περίπτωση της χώρας μου να έχουμε 20 εθνικά στατηγικά σχέδια. Αυτό συνεπιφέρει άμεσο κίνδυνο που είναι τεράστιος, συγχρηματοδοτήσεως όλης της ΚΑΠ διότι πώς θα πούμε ότι στο δεύτερο πυλώνα συγχρηματοδοτούμε 50% και τα υπόλοιπα μένουν 100% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν είναι εθνικό σχέδιο θα είναι όλα στη συγχρηματοδότηση. Να μην μιλήσουμε μετά για τους κινδύνους τρέβλωσης, διότι αναφυσβήτητα ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα πετύχουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί τρόποι. Σε κάποιες χώρες εκεί θα βασιστούν στη ζωοτεχνία, άλλοι στην παραγωγή, ε, την οποροκυπευτική θα υπάρχουν στρεβλώσεις. Διότι ακριβώς αυτό που γραμμίσαμε αρνητικά για την παρούσα ΚΑΠ είναι αυτό. Θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το περιεχόμενο. Βέβαια, οι υποθέσει είναι πολύ καλέ, ιδεώδη κόσμο. Θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα ιδεωδώ. Θα υπήρχαν και θετικέ πτυχέ. Αλλά στην πραγματικότητα, μετά στην πρακτική εφαρμογή, θα αντιμετωπίσουμε διαφόρου σημαντικού κινδύνου επανεθνικοποίησης, κινδύνου συγχρηματοδοτήσεως, κινδύνου ε, χρηματοπιστωτικών διοθώσεων. Διότι αν τα κράτη-μέλη δεν πετύχουν μετά τους target, θα υπάρχουν κυρώσει. Και εγώ ήδη φαντάζομαι χώρε με μεγάλη περιφερειοποίηση που έχουν προβλήματα τεράστια ε, να πρέπει να διαχειριστούν τις ε, κυρώσεις στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού. ευτυχώς έχουμε το χρόνο, διότι αυτή η θητεία και το λέω στους συναδέλφους, αυτή η θητεία δεν θα μπορέσει να εγκρίνει τίποτα. Διότι υπόθηκε σαφέ, σαφώς με την Omnibus κάναμε έξοχη δουλειά, ευχαριστώ τον Ρούλοφ Μάιερ γι' αυτό, αλλά χρειαστήκαμε 14 μήνες. Πώς να διανοηθούμε να κάνουμε τα ρύθμιση τόσο περίπλοκη, τόσο διαφρομένη που αλλάζει εντελώ την αρχική βάση και το πλαίσιο σε λιγότερο από 1,5 χρόνο. Ευχαριστώ. Ε, εγώ νομίζω ότι ε, η, η ζωή είναι πιο επίκης. Θα δούμε όμως ε, πώς θα εφαρμόσουν όλα αυτά οι γεωργοί. Και οι στόχοι είναι κάπως ε, θεϊκές ε, επιθυμίες. Κύριε Κάντεμπαχ. Αν ήταν στόχοι τόσο συγκεκριμένοι, δεν θα αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα μια έκθεση δηλαδή του ελεκτικού συνεδρίου σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Ε, είναι ακριβώς αυτό που δεν έχει διαμορφωθεί σαφές ε, στους στόχους αυτούς και γι' αυτό λοιπόν είναι, είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε κατά πόσον ε, με τα χρήματα που δαπανάμε πετυχαίνουμε αυτή την προστεθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Υπογραμμίζω λοιπόν αυτά που είπαν οι συνάδελφοι Χόισλεν και Δεκάστρο σε ό,τι αφορά τον παράγοντα του πράσινου προσανατολισμού, το πώ θα προσμετράτε στο μέλλον και πώ θα χρηματοδοτείτε αντίστοιχα. Γιατί προχθέ από αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβα ότι αυτά τα μέτρα για το πρασινίσμα δεν είναι τόσο μέθοδος ε, καθοδήγησης ε, προς τη βιώσιμη αγροτική πολιτική, αλλά απλά δεν θέλει δηλαδή να πετύχει αλλαγή της γεωργίας με, το, με τη δαπάνη αυτή. Εγώ δεν καταλαβαίνω έτσι την πράσινη προσέγγιση, τον πράσινο προσανατολισμό. Έχουμε το performance orientation σε ό,τι αφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεκτική ομάδα δικτών για τις απαραίτητες προδιαγραφές για τις επιδοήσεις και για τις στόχους σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την ΚΟΑ. Από πολλές εκθέσεις έχουμε διαπιστώσει ότι όλοι αυτοί οι στόχοι και αυτοί οι δείκτες δεν υφίστανται ουσιαστικά προκειμένου να μπορέσουμε να τους διαπιστώσουμε και να τους αναπτύξουμε. Ε, μα πώς φανταζόμαστε ότι στον περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας θα καταφέρουμε να ορίσουμε σωστούς δείκτες για να μπορέσουμε με προσμετρήσιμο τρόπο να αποδείξουμε ότι έχουμε πετύχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια να αναπτύξουμε περαιτέρω εθνικούς ε, δείκτες σε επίπεδο κρατών μελών, σε 27 κράτη-μέλη. Τι να σας πω, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα το πετύχουμε αυτό στο περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχουμε. Και πολύ φοβάμαι ότι και η επόμενη έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου τα ίδια συμπεράσματα θα εξαγαγεί. Και πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι που θέλουμε. Ο κύριος Κολομπιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή... Παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια απλούστευση των διαδικασιών, αλλά εγώ τελικά βλέπω μια ένα πολλαπλασιασμό των ε, προδιαγραφών και είναι η άποψη των γεωργών. Ε, για τους γεωργούς προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Όσον αφορά τη μείωση που ανακοινώνεται για τον προπολογισμό για την ΚΑΠ, πολλοί δρόμοι ε, τελικά υπονομεύουν τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ και ε, για τις ενισχύσεις. Αν μπορεί να βελτιωθεί ο τρόπος καταβολής των πληρωμών των ενισχύσεων, θα πρέπει να δούμε ότι οι πρώτερες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ δημιουργήσαν τη βασική δυσλειτουργία και τα προβλήματα δηλαδή την αποσύνδεση η οποία ε, στηρίζει την έκταση ένα της εργασίας και το πρασίνισμα που κατά την άποψή μας είναι κάτι αναποτελεσματικό και δαπανηρό. και να συνοψίσω, λίγο πολύ τα ίδια πράγματα είναι. Δηλαδή, ενώ σαμποτάρανε τον πρώτο πυλώνα, μας ζητούν τώρα να μειωθεί αυτός ο πυλώνας και να καταργηθεί. Υπονομεύονται οι άμεσες πληρωμές. Ενώ τίποτα δεν ανακοινώνεται ότι ολοκληρώνεται, ε, περνάει η κρίση που έπληξε τους καλλιεργητέ κατα, καταδικάζει τελικά αυτούς που απομένουν στη χρεοκοπία. Αυτή που είτε είναι κανεί κατά ή υπέρ τη ε, των άμεσων πληρωμών, είναι πραγματικότητα. Πρέπει να γνωρίσουμε. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση κάνουν τι επιλογέ και κατά τη μελλοντική μεταρρύθμιση, να ξέρουμε ποιε είναι οι συνέπειε αυτών που προτείνουμε. Ευχαριστώ. Ο Δαντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή Ούτε μια φορά δεν χρησιμοποίησατε τη λέξη οικονομία. Η ΚΑΠ καταρχάς είναι μια οικονομική πολιτική. Για μία ακόμη φορά θα πρέπει να υπομειώσουμε το άρθρο 39 των συνθήκων που στο σημείο Β μας λέει ότι η ΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίζει επίπεδο δίκαιο διαβίωση στον γεωρικό κόσμο μέσω μια στήριξη του ατομικού εισοδήματο εκείνων που εργάζονται στον αγροτικό τομέα. Να υπενθυμίσουμε το σημείο Γ να σταθεροποιεί τη αγορά θα πρέπει να θυμίσουμε και το σημείο ε να εξασφαλίζεται η λογική τιμή όσον αφορά τι παραδόσει των προϊόντων στου καταναλωτέ. Προτείνεται ένα νέο μοντέλο για την εφαρμογή των μέτρων, μια αρχιτεκτονική ακόμα πιο πράσινη. Τώρα, όσον αφορά το νέο μοντέλο τη εφαρμογή των στόχων, βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει, υπάρχει κάτι ζωσπαστικό. Ε, θέλουμε μία απλούστευση, αλλά η απλούστευση είναι για τι υπηρεσίε σα. Για να απαντήσουμε φιώ στα διάφορα ερωτήματα που ετέθησαν, ε, για να, για να μειωθεί, θέλετε να μειώσετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις θέσεις εργασίας και, και το μεταφέρετε σε επίπεδο 100 μελών. Εγώ σας προτείνω κάτι απλό. Δώστε μας ένα στρατηγικό σχέδιο που, μοντέλο που θα μας δείχνει λεπτο, ε, λεπτομερώς τι περιθώρια λιγμών έχουν τα κράτη-μέλη και τι αυτή η περιπτώση. Αν συμφωνήσουμε θα υπογράψουμε τελικά ήσυχη όσον αφορά αυτό που κάνουμε, σίγουρα αυτό που κάνουμε. Με αυτό που μας προτείνεται όμως, η αρχιτεκτονική είναι τέλεια, δεν έχουμε καμία διευκρίνηση όσον αφορά το περιεχόμενο. Ποιος θα αξιολογήσει αυτά τα σχέδια, ποιος ε, θα, θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας θα είναι η μόνη ή θα υπάρχουν διάφοροι ε, οι οποίοι θα θέλουν να πάρουν χρήματα από τον προπολογισμό της ΚΑΠ. Δεν έχουμε καμία πληροφορία, κανένα όραμα. Ποιος θα είναι ο ρόλος του συνομοθέτου, των συνομοθετών όσον αφορά τον έλεγχο των ε, σχεδίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το κάνει αυτό. Αλλά με αυτό το μηχανισμό τελικά αφήνεται εκτός τους ε, συνομοθέτες και δεν μπορούν να εκτελέσουν την αποστολή τους. Λοιπόν, μπορείτε, ε, εάν μας δώσετε ένα υπόδειγμα σχεδίου θα το μελετήσουν προσεκτικότατα όσον αφορά τα μέτρα της πράσινης αρχιτεκτονικής φοβούμε μετά τις εξηγήσεις που μας δώσατε ότι ξεκινάμε για 70% 100% υπεραιρεσιμότητας αν θέλετε. Περιμένουν κάτι άλλο οι Γεωργοί από εμά. Περιμένουν να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα ένα πλαίσιο που τους επιτρέπει τελικά να έχουν ένα εισόδημα. Ο κύριος ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Ντόρφμαν για το σχέδιο έκθεση που θα αποτελέσει πολύ καλή βάση εργασία για τι περαιτέρω συζητήσει. Κύριε Μέγκελε, και εγώ άκουσα με προσοχή την ομιλία σα και, και πιστεύω ότι ουσιαστικά είναι η απόφαση της αποτυχίας ε, πεντε, ε, ΚΑΠ. Γιατί όπως είπαμε, η πρωταρχική λειτουργία της είναι η εξασφάλιση της γεωργίας και του γεωργικού εισοδήματος. Και οι αγορές είναι πάρα πολύ ασθενείς, οπότε έχουμε φοβερό, φοβερές ανησυχίες και προβληματισμό. Επίσης, ε, για τους νέους γεωργούς, ε, η αλλαγή της μεθόδου δεν νομίζω ότι θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε την πρόκληση της διασφάλισης του γεωργικού εισοδήματος, ε, της σύνδεσης ε, ε, του γεωργού με το τρόφιμο, με την υγεία, με το περιβάλλον, που είναι δημόσια αγαθά. Είναι σημαντικοί οι στόχοι και ενδιαφέροντες, αλλά νομίζω ότι η ευθύνη σε κοινοτικό επίπεδο είναι να είμαστε πιο κοντά στους στόχους και το γεγονός ότι μιλούμε για εθνικά στρατηγικά σχέδια. Καλύτερα να μιλάμε για, για εθνικά επιχειρησιακά σχέδια και όχι στρατηγικά. Είπατε ότι ο προσανατολισμός στηρίζεται σε κοινού ευρωπαϊκούς στόχους που θα συμπληρώνονται από πιο συγκεκριμένου εθνικού στόχου. Πώ είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε έτσι μια συνοχή και μια αξιοπιστία για την υλοποίηση των στόχων. πώ θα γίνει η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων. Και εγώ ανησυχώ τα μάλα από το ρόλο που δίνετε στην πρότασή σας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικώ στους συνομοθέτες. Ε, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ερωτήματα σήμερα, πολλό δε μάλλον που είναι πολύ στενές ε, οι προθεσμίες για τη μεταρρύθμιση. Πάντως, το μείζον ζήτημα είναι μια ανοιχτή αγορά σε διεθνέ επίπεδο και η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει με οικονομικά εργαλεία να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη της ανοιχτής αγοράς παγκοσμίω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Τόρφμαν για την ε, ταχύτητα και τη διαφάνεια με την οποία εργάστηκε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ομιλία της, για την παρουσίασή της και για τη διαμόρφωση του οικολογικού προσανατολισμού και της αιρεσιμότητας. Ε, κάποιο, κάποιες ενδείξεις γίνεται για τα γενικά, αλλά ελάχιστα για τα συγκεκριμένα. Ποιε είναι οι συνέπειε αυτή τη νέα πρόταση για του αγρότε και τι εθνικέ διοικήσει. Λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση, ο αντίκτυπο των νέων προτάσεων στου αγρότε και τι εθνικέ διοικήσει. Είπατε ότι ε, ο πρώτος πυλώνας της ΚΑΠ θα, περιληφθεί στην ίδια, στον ίδιο τρόπο διακυβέρνηση με τα διαφορετικά ταμεία, δηλαδή ε, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και τις άμεσες ενισχύσεις των πρώτο πυλώνα θα συνδυάσετε με το δεύτερο πυλώνα ε, τη, την αγροτική ανάπτυξη. Τι ε, χέγγια θα δώσετε για την συγχρηματοδότηση του πρώτου πυλώνα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πληρωμών. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγγείλει ότι θα συνδέσει ε, το θέμα αυτό με τους δικαιούχους και θα κάνει έναν έλεγχο με βάση τα αποτελέσματα, πώς θα εξασφαλίσετε ότι το αποτέλεσμα χ γεωργικών εκμεταλλεύσεων ε, βιολογικής γεωργίας ανταποκρίνονται πραγματικά στη βιολογική γεωργία. Πώς θα πραγματοποιήσετε αυτούς τους ελέγχους. Ευχαριστώ. Κυρία Καλνιέτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Ντόρφμα για το σχέδιο έκθεσης. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ήταν μόνο μερικώς επιτυχής. Οι προτάσεις που έχουμε σήμερα μπροστά μας θα έλεγα ότι προκαλούν σύγχυση. Δεν απλοποιούν, αλλά περιπλέκουν περαιτέρω. Να σας Επίσης, ε, να σας προειδοποιήσω και ότι θα είναι πραγματικά παράδεκτο να υπάρχει μείωση και αφαίρεση της χρηματοδότησης της εθνικής σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση προϊόντων και γεωργικών πρακτικών για τους ε, γεωργούς στη χώρα μου. Το θέμα είναι η σύγκληση των άμεσων ενισχύσεων, γιατί οι άμεσες ενισχύσεις για τη Βαλτική είναι οι χαμηλότερες από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ χαμηλότερες του μέσου όρου. Αυτό δεν είναι βιώσιμο, δεδομένου του ότι οι γεωργοί μας αντιμετωπίζουν το ίδιο κόστος, τις ίδια έξοδα, τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και όλοι οι υπόλοιποι εργοδότες στην Ευρώπη. Επίσης, να τονίσω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η δομή με τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές ε, για το δεύτερο πυλώνα, είναι πολύ πιο υψηλέ για τα κράτη-μέλη και ότι αυτό θεωρητικά θεωρείται ότι δικαιολογεί τις χαμηλότερες άμεσες ενισχύσεις. Αυτή είναι μια πλάνη, δεν ισχύει και έχει αποδεχτεί επανειλημμένα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω ίση κατανομή των ε, πόρων και στους δύο πυλώνες της ΚΑΠ. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Αναπτύξης της Υπέθρου θα πρέπει να δημιουργεί ίσους όρους του αγωνισμού σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την ανάπτυξη. Αυτό λείπει ακόμα γιατί είναι χαμηλό το επίπεδο του κατακεφαλής ε, εισοδήματος. Άρα, συνολικά, θα ήθελα να αναγνωρίσω ότι η τρέχουσα πρόταση και οι τρέχουσες προτάσεις μάλλον προκαλών σύγχυση αποτελούν ωστόσο μια πλατφόρμα για να σχεδιάσουμε μια πιο σωστή και σύγχρονη ΚΑΠ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Χάζεκαμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει και εξοδεύει λεφτά ε, σαν νερό. Έχουν ανοίξει οι βρύσες και 40% του ευρωπαϊκού προπολογισμού χάνονται σε επιδοτήσεις αγροτικές. Προσβλέπουμε στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά Πρωτού συνεχίσει το τρένο των επιδοτήσεων, θα ήθελα να κοιτάξω λίγο τι έχει γίνει ως τώρα και να κάνω μια σύντομη περισυλλογή. Η Ολλανδία έλαβε άμα, 725 εκατομμύρια πέρσι σε αγροτικέ επιδοτήσει. και αυτό ουσιαστικά ωφέλησε τι μεγάλε οργανώσει και τα σούπερ μάρκετ. Αυτοί πήραν τα μεγάλα ποσά. Είναι ντροπή και όνειρο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύουμε και σπαταλάμε ε, προϊόντα για, ε, χρήματα για προϊόντα που είναι αντίθετα στην ευημερία των ζώων για τις μεγάλες ε, μεγάλες κλίμακες αποθηκεύσεις ε, κρέατος. Υπάρχουν υποτίθεται κάποια μέτρα για το πρασίνισμα, τα οποία όμως δεν έχουν οποιαδήποτε αντίκτυπο για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η ενίσχυση για την πράσινη προσανατολισμό αποτελεί μια ενίσχυση εισοδήματο και τίποτα παραπάνω. Πώ θα τα εξηγήσουμε αυτά, Πρόεδρε, στα φορολογούμενα, ότι με τέτοιε μεγάλε δαπάνε στην Ευρώπη ε, και εκατομμύρια ζώα υποφέρουν ε, στην κτηνοτροφία. Και ουσιαστικά ο τρόπος ε, με τον οποίο δουλεύουμε μολύνει τα ύδατα μας, χαλάει τη βιοπικιλότητα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να το εξηγήσουμε αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συγητής συνεχίζουν το χαβά τους θα πρέπει, Πρόεδρε, να γίνει μια δραστική αλλαγή, γιατί ο πλανήτης μας υποφέρει και θα καταρρεύσει από την έντονη εκτροφή και καλλιεργία. Θα πρέπει να υπάρξει ζωσπαστική αλλαγή στον τρόπο ε, καλλιεργίας και εκτροφής. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε και διαφορετικά το σύστημα τετροφής μας να καταργήσουμε τις αγροτικές επιδοτήσεις και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να καταργηθεί ολοσχερός το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων. Ευχαριστώ κύριο Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε. Και να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει, βεβαίως και αλλάζει και σε μια χρονική στιγμή όπου καταρτίζουμε ένα κοινό σχέδιο για την άμυνα και την ασφάλεια. τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα Ασφάλεια τροφίμων. Για μένα το πιο μεγάλο και το πιο βασικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για μένα αλλά και για τον κόσμο που εκπροσωπώ είναι να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια τροφίμων, μια ενιαία αγορά για τα προϊόντα μας τα οποία να είναι ίδιας ποιότητας. Εκεί λοιπόν υποστηρίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε άλλους τομείς δεν θα την υποστηρίζα. Να πω λοιπόν ότι θα πρέπει να, όχι να περικόψουμε τον προπολογισμό μας, αλλά να αυξήσουμε τον προπολογισμό μας για να έχουμε πιο πολλά υπεύθυνα έργα. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά το πώς εφαρμόζονται και πώς χορηγούνται τα χρήματα αυτά, γιατί θεωρητικά ακούγεται πάρα πολύ καλά το, πρόγραμμα, αλλά στην πράξη πώς διαμορφώνεται. Το μοντέλο του, του δεύτερου πυλώνα έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου ο κόσμος τριμώχνεται έξω από το γραφείο μου και έξω από το γραφείο άλλων βουλευτών για να μιλήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα είναι ανοιχτή για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά τελικά μας, ε, στέλνει, τους στο σπίτι τους χωρίς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά και είμαστε οικογένεια και ο μπαμπάς μας στέλνει στη μαμά και η μαμά στον μπαμπά. Το είπαμε στο σκύλο μας και ο σκύλος στην ουρά του. Τι έγινε λοιπόν, τι θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί με την τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Σωστή σύγκληση. Αν θέλουμε να γίνει επιτέλους αυτή η σωστή σύγκληση, θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Στη χώρα μου κάποιοι άνθρωποι παίρνουν 1000 ευρώ ανά εκτάριο και οι γείτονές τους μπορεί να παίρνουν μόνο 100 ευρώ ανά εκτάριο. Μπορεί να παίρνουν 30 ευρώ ανά εκτάριο για πράσινο προσανατολισμό και οι γείτονές τους να παίρνουν 300 και 400 ευρώ για τον ίδιο σκοπό. Όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν. Αν υπάρξει δικαιοσύνη, μπορεί να υπάρξει μεγάλη αλλαγή για την ε, οικονομία της υπαίθρου και όλο αυτό να επηρεάσει με τη σειρά του την, ε, τις, τα μικρά αγροκτήματα. Το είπατε κύριε Ντόρφμαν και ξέρω ότι το εννοείτε ότι όλα αυτά θα πρέπει να στραφούν τελικά και να διοχετευτούν στι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και θα πρέπει να γίνουν υπολογισμοί βάσει ιστορικών ε, κριτηριών. Τότε μόνο μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Γιατί δεν βλέπουμε πραγματικά αυτά τα χρήματα να φτάνουν στο, στον κόσμο, στη συνήπεθρο. Αυτά τα χρήματα τελικά καταλήγουν σε δυτικά τζετ, σε κοσμήματα του στέματος σε κάποιες περιπτώσεις ε, Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη τέτοια επιρροή. Ναι, σίγουρα η επιστηστική ασφάλεια είναι αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής έννοιας της ασφάλειας. Ας μην το ξεχνάμε. Ο κύριος Λίτς. Σας ευχαριστώ και καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Ντόρφμαν γιατί θεωρώ ότι η έκθεση του είναι πολύ επιτυχημένη αποτελεί μια καλή βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις μας ε, επί της έκθεσης αυτής. Και την διαπίστωση επίσης ότι αν ε, έχουμε ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκούς πόρους και θέλουμε να τους ελέγχουμε, πρέπει να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Έχω δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνω αν σωστά κατάλαβα. Σε ό,τι αφορά το delivery model, το μοντέλο παροχής, ε. στους ε, δύο πυλώνες της ΚΑΠ, έχετε υπόψη σας ε, η διαμόρφωση των λειτουργικών προγραμμάτων να γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών και μόνο. Εγώ είμαι από ένα μεγάλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχουμε ομοσπονδιακό σύστημα με ομοσπονδα κρατήδια. Μεγέθους ε, εξίσου μεγάλου όσο κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρωτώ, λοιπόν, θα πετύχουμε μείωση της γραφειοκρατίας. Αν στο δεύτερο πυλώνα των, της ΚΑΠ έχουν ορμοδιότητα μόνο τα κράτη-μέλη και έτσι ουσιαστικά αφαιρέσουμε την επικουρικότητα. Έτσι κατάλαβα ότι είπατε ή μήπως κατάλαβα κάτι λάθος. Κατά δεύτερον, σε σχέση με αυτά που είπε και ο συναδέλφος Νταντά. Συμφωνώ. Αν σωστά κατάλαβα, τα μέσα για το πρασίνισμα θα πρέπει να μπουν στον δεύτερο πυλώνα. Αλλά η πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να τευρυνθεί. Σημαντικά. Θα ήθελα να έχω πιο πολλές λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό. Το ερώτημα σε ό,τι αφορά επίσης ε, τη σύνδεση πρώτου με δεύτερο πυλώνα. Πώς θα γίνει αυτό. Και πώς θα αντιμορφωθεί η συγχρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τη γεωργική περιβαλλοντική πολιτική στο δεύτερο πυλώνα. Αυτό θα αποτελούσε μεγάλη πρόκληση για κάποια κρατημέλη. Κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μ' αρέσει η ιδέα που εστιαζόμεθα στα επιτεύγματα αυτά κάθε αυτά και όχι τον τρόπο επιτεύξεως. Πρέπει να εκταθεί ο κατάλογος να συμπεριλαμβάνουμε τη συντηρητική γεωργία, τα σχέδια όσον αφορά τις ε, διάφορες ε, θρεπτικές ουσίες κλπ. Είναι βάση αυτά που προτείνεται και μετά οι γεωργοί πρέπει να κάνουν περισσότερα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο από την παρουσίαση. Μετά οι γεωργοί, είτε είναι οικογενειακέ εκμεταλλεύσει, μεσαίου μεγέθου, μικρέ ή μεγάλε εκμεταλλεύσει, χρειάζονται βεβαιότητα. Είναι επιχειρήσει. Και δεν βλέπω από την παρουσίαση να υπάρχει βεβαιότητα σήμερα. Δεν κατανοώ ακόμα κατά πόσο μιλάμε για υποστήριξη με βάση την έκταση και τη γη του πυλώνα 1, κατά αποκοπήν αναεκτάριο πληρωμές του πυλώνα 1, αν όλες αυτές οι πληρωμές το 100% θα προϋποθέτει συμπληρωματικές ε, προϋποθέσεις των περιβάλλων. Πώς θα πληρούνται οι προϋποθέσεις. Μετά το άλλο, η συνοχή. Στην Ιρλανδία, παραδείγματο χάρη. Έχουμε ε, διάφορα βαλτόδια εδάφη, είναι υδροβιότοποι. Για να συμμορφωθούμε με τη σωστή γεωργία και περιβαλλοντικές συνθήκες, οι γεωργοί ε, ψεκάζουν αυτές τις περιοχές και μπαίνει στο νερό. Ψεκάζουν τα φυτά, μπαίνει στο νερό αυτό που ψεκάζουν και μολύνουν τα ύδατα. Ε, θα ήθελα να υπάρχει συνοχή, να πληρώνονται για τους βιοτόπους που υπάρχουν στις εκμεταλλεύσεις τους. Αυτό είναι το βασικό μου μήνυμα, να μην πληρώνονται να καταστρέφουν ένα βιότοπο, να τον καταστρέφουν και να φυτεύουν κάτι για να ενταχθούν τελικά σε κάποιο πρόγραμμα. Μετά μπορεί να καθορίσει κανείς ε, τι είναι η δικαιοσύνη, τι εννοούμε με δικαιοσύνη διότι αναφέρεται επανειλημμένα εδώ και αλλού. Να είμαστε δίκαιοι απέναντι στον κάθε Γιωργό, απέναντι στην εκμετάλλευση, απέναντι στην οικογένεια, απέναντι στην κοινωνία. Στο συλλογικό μας νου, ποιος είναι ο ορισμός του δίκαιου, ένα δίκαιο που θα λειτουργεί για μια πανευρωπαϊκή κοινή αγροτική πολιτική. Πόσο ο κύριος Βογκόβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον Χέρμπερτ Ντόρφμαν για το σχέδιο εκθεσής του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί απλούστευσης και τα λοιπά. Καταρχήν, ο κυριότερος εχθρό τη απλούστευσης είναι οι ρηξικέλευθες αλλαγέ, οι νέε προσεγγίσει, η έλλειψη σαφήνεια, οι καθυστερήσει και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η εχθρή της απλούστευσης. Σχεδόν φτάσαμε άνοιξη το 2018 και νομίζω θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα με αυτά της πολιτικής συνοχής. Και εκεί είχαμε κάποιες ε, σημαντικές επαναστατικές αλλαγές, αλλά ελάχιστη σαφήνεια και ήδη έχουμε μείνει πίσω, ήδη υπάρχει καθυστέρηση, οπότε πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Ε, δεν έχουμε αρκετά κονδύλια για επιστηστική ασφάλεια, δεν έχουμε αρκετά κονδύλια για τη γεωργία. Τώρα, βέβαια, ενώ δεν έχουμε καν 1% για τη γεωργία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αφιερώνουμε 2% για τις αμυντικές δαπάνες, για το ΝΑΤΟ. Η πιστιστική πολιτική και η αγροτική πολιτική είναι και κοινωνικές πολιτικές ταυτόχρονα. Γιατί οι καταναλωτές αφιερώνουν το 50-60% του προπολογισμού τους για τα τρόφιμα. Απ' την άλλη έχουμε αγρότες που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα προβλήματα. Το δείχνουν ξεκάθαρα οι στατιστικές. Και φυσικά θα πρέπει να στηρίξουμε τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, να διαφυλάξουμε τις γεωρικές εκμεταλλεύσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τους ε, γεωργούς που ξεκινούν γεωργική δραστηριότητα για να έχουν ε, προσδοκίες σε ένα καλό μέλλον και φυσικά καλύτερο, περισσότερο greening και πιο ακριβωδική κατανομή μεταξύ των χωρών και μεταξύ των γεωργών αλλά και στο θέμα των διαστάσεων και του μεγέθους. Χρειαζόμαστε πρακτικές λύσεις. Και δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Τώρα για τον οικολογικό προσανατολισμό, το greening, πιστεύω ότι με την πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις καλές πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές για το περιβάλλον και τους πολίτες. Και φυσικά πάλι δίκαιη κατανομή και να ενθαρρύνουμε τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία και καινοτομία και νέα γνώση με την ψηφιοποίηση για να φτάσουμε και στα έξυπνα χωριά και σε μια ζωντανή ε, ύπεθρο στην οποία θα διαβιούν όλες οι γενιές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστερημένος. Έπρεπε να ψηφίσω άλλη επιτροπή. Θα ήθελα να ήμουν παρόν κατά τη διάρκεια της συζητήσεως. Υπάρχει αοριστολογία εδώ. Μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, μεσές εκμεταλλεύσεις, μικρές εκμεταλλεύσεις, λέμε εδώ. Ποιος αποφασίζει περί μεγάλης εκμεταλλεύσεως και από τρεις μεριές το βλέπει κανείς. Έκταση, μετά συγκρίνεις 5.000 ορεινό, ορεινή εκμετάλλευση με 100 στη Σκοτία, με 100 στο νοτιοανατολικό και εκεί ε, μικρότερη έκταση μπορεί να παράγει πολύ περισσότερα προϊόντα από μεγαλύτερη έκταση αλλού. Μπορεί να δει κανείς τζίρο, παραγωγή, αριθμό εργαζομένων. Από τη στιγμή που ακολουθεί αυτή την προσέγγιση, που προσπαθεί να καθορίσει τι είναι μεγάλο και τι δεν είναι μεγάλο, κυρίω εάν ταξιδεύσει στην Ήπειρο και αυτό που είναι μια μικρή εκμετάλλευση στη Βρετανία μπορεί να θεωρηθεί αρκετά μεγάλη εκμετάλλευση κάπου στην Ανατολική Ευρώπη θα ήταν πολύ ευκολότερο κατά την απόψή μου απλώς να βάλετε ένα ανώτατο όριο για την πληρωμή σε κάποιο επίπεδο και να ξεμπερδεύετε. Αν δεν αρέσει αυτό, αν δεν αρέσει αυτό σε κάποιον να πει στο γιο του, κοίτα, έχεις μισό από αυτό, ε, τώρα είναι δύο εκμεταλλεύσεις και εσύ και εγώ μπορούμε να αξιώσουμε πληρωμές, το μοιραζόμαστε, το ένα το κάνουμε δύο και μοιραζόμαστε. Όσον αφορά του ορισμούς, δεν αναφέρεται εδώ στο έγγραφο, αλλά πολύ συχνά από τους πρασίνους αναφέρεται η βιομηχανική εκμετάλλευση, εκμετάλλευση εργοστάσιο, factory farm. Τι είναι αυτό. Δηλαδή, αν βάλεις, αν πας ένα πολύ παραπάνω, παραδείγματος χάρη, ε, μπορείς, ε, να προσ... Ε, ε, μπορείς να βάλεις ένα, ένα χείρο παραπάνω, ένα πολύ παραπάνω στην εκμετάλλευση και να αλλάξεις κλίμακα. Ε, τι εννοούν τελικά με την εκμετάλλευση βιομηχανικής ε, κλίμακας. Πρέπει να λειτουργούν εντός καθορισμένων κλιματολογικών στόχων. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Τι στο καλό σημαίνει αυτό. Το συζήτησα εκτενώς. Αλλά άμα ακολουθήσει το δρόμο πρέπει να πεις, πρέπει να μειώσεις διοξείδιο του άνθρακος, ε, κατά τα οξύδια του αζότου, ε, το, το άζωτο κατά άλλη ποσότητα. Αλλά ποιο είναι αυτό είναι καλό να αναφέρεις αυτά, δεν θα κάνει διαφορά τελικά, αλλά είναι ένας διοικητικός εφιάλτης όλοι αυτοί οι ορισμοί εδώ. Κύριε Γιάρα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη, χαίρομαι πάντα που έχει αμφιβολήσει ο κύριος Σεκ για τη συνέχιση της γεωργικής πολιτικής, αλλά, αλλά τουλάχιστον να μείνει μαζί μας, άμα τον ενδιαφέρει να την διαμορφώσει. Δεύτερη παρατήρηση. για τον πρόεδρο. Με τις δέκα εντολές, ε, ο Αλμπερτές ε, μου είπε ότι οι δέκα εντολές αυτές ε, λειτουργήσαν γιατί δεν ήταν νομικοί στην κατάρτιση τους, δεν συμμετείχαν. Τρίτη παρατηρήση. για τον κύριο Μπόκοβιτς. Ε, δεν ξέρω αν έκανα λάθος, αλλά νομίζω ότι η αγροτική πολιτική δεν είναι κοινωνική πολιτική, είναι πολιτική ασφαλείας η πολιτική αυτή. Γιατί το θέμα είναι να, υπάρξει, να υπάρξουν τρόφιμα για τον κόσμο στην Ευρώπη, άρα δεν βλέπω γιατί είναι κοινωνική πολιτική. Το... Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Εγώ θέλω να μας απαντήσει ο συνάδελφος Γκλίντσε Δεύτερη παρατήρηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντόρφμαν για την έκθεσή σου. Για μένα η έκθεση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει την γέφυρα μεταξύ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πρακτικής εφαρμογής, γιατί για αυτήν είμαστε υπεύθυνοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθυστέρησα να έρθω γιατί είχα και συνάντηση συντονιστών, αλλά δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει την εντύπωση ότι φοβούμαστε την ε, απολευθέρωση τέτοιων συστημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν μας έχει δώσει πάρα πολλές προδιαγραφές και αυτό μας έχει φοβήσει. Τώρα ακολουθεί μια διαφορετική οδό και νομίζω ότι θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία αυτή. Και αυτό κάνει και ο κ. Ντόρφμαν ε, στην έκθεση του φυσικά. Το θέμα δεν είναι μόνο η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, κρατών μελών. Το θέμα είναι να μπει στο επίκεντρο ο αγρότη και αυτό νομίζω δεν προσθέτει αρκετά στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επόμενη ερώτηση. Θα υπάρξουν μεταβατικέ περίοδοι, γιατί το τόνισαν διάφοροι συναδελφοί ότι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους ε, στη χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε ορίσει, θα χρειαστούν μεταβατικές περίοδοι. Κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Τα αποτελέσματα της προσέγγισης αυτής είναι ένα λεπτό ζήτημα για την κοινή πολιτική. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα θέμα που δεν ε, αναφέρθηκε αρκετά. Τη θέση των ε, αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού, στην αλυσίδα τροφίμων. Βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι έχουμε μια οικονομία της αγοράς και πολλά από τα προβλήματα του χαμηλού γεωργικού εισοδήματος οφείλονται στην πολύ ασθενή, αδύναμη θέση των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Επίσης, στην επόμενη ε, περίοδο χρηματοδοτική θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα συνδυασμού των δύο πυλώνων και σίγουρα ε, τα κράτη-μέλη να έχουν τον περισσότερο λόγο για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του πρώτου πυλώνα. Σε ό,τι αφορά τις διάφορες θέσεις των κρατών μελών για τα διάφορα επίπεδα άμεσων ενισχύσεων, η κατάσταση ιδεοδός θα ήταν όταν ξεκινήσουμε τη συζήτηση κατά το 2020 να έχουμε λιάνει ήδη τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών για να μην υπάρχουν τέτοιες διαφορές μεταξύ τους. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερα στη χθεσινή έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Πιστεύω ότι αν δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να κάνουμε έναν απολογισμό των πολιτικών μας και να δούμε πώς εφαρμόστηκαν στην πράξη, πώς είναι δυνατόν να σχεδιάσουμε νέες πολιτικές σε ό,τι αφορά τις άλλες πτυχές της κοινή γεωργικής πολιτικής, θα πρέπει και εκεί να αξιολογήσουμε το πώς λειτουργήσαν τα μέτρα μας για να αποφασίσουμε τι μέτρα χρειάζονται για το μέλλον. Μάλιστα, δύο ακόμη συναδέλφους έχω στον κατάλογο. Τον κύριο Ντες πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους, λοιπόν, της μεγαλύτερης ομάδας του Κοινοβουλίου, πρέπει να πω ότι συνήθως έχουμε κάποιες προτεραιότητες. Ήθελα να περιμένω μέχρι το τέλος της συζητήσεως. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση και ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προβληματισμό που έκανε όσον αφορά το θέμα αυτό. Δεν είχαμε δει κάποια συγκεκριμένη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον τρόπο, με τον... Ε, μάλλον προτείνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς βελτιώνουμε συνήθως το κείμενο. Λοιπόν, με την τρέχουσα ΚΑΠ ε, έχουμε πολλά περιθώρια για τα κράτη-μέλη ε, έχουμε πολλά μοσπονδακρατήδια κρατήδια στην Ευρωπαϊκή, στη Γερμανία. Έχουμε 12 εκατομμύρια κατοίκους εμείς στη Βαβαρία. Έχουμε πολλές εγγελικές εκμεταλλεύσεις. Είδα τα στατιστικά στοιχεία. Μόνο 5% από τις εκμεταλλεύσεις στη Βαυαρία έχουν πάνω από 100 εκτάρια. 50% έχουν μέχρι 20 εκτάρια. Άρα έχουμε πολύ μικρές υποδομές στη Βαβαρία. Βλέποντας τα στοιχεία οι Βαβαροί Γεωργοί παίρνουν 500 εκατομμύρια ευρώ ε, στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα και ένα δις στο δεύτερο πυλώνα, διότι η Βαβαρία χρησιμοποιεί τα προγράμματα και μας κοστίζει ελάχιστα. Από τα 100 ευρώ που πληρώνουμε στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα, τα 20 ευρώ προέρχονται από τη Βαβαρία, 30 από το Βερολίνο και 50 ευρώ από τις Βρυξέλλες. Διαπιστώνω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη δεν αξιοποιούν αυτέ τι ευκαιρίε και τα χρήματα του δεύτερου πυλώνα ωφελούν ε, τι ε, οικογενειακέ επιχειρήσει. Πάνω από 60% των επιχειρήσεων στην Βαυαρία είναι σε ε, προγράμματα πράσινου προσανατολισμού και παίρνουν επι, ενισχύσεις. ενισχύσει. Σα ε, παρακαλώ λοιπόν να διαβάσετε την έκθεση του κ. Μαρτίν που αναφέρει και υπολογίζει τέτοια ποσά. Γιατί, Γιατί θέλουμε να δούμε ποια... Υποτίθεται ότι θέλουμε να αφαιρέσουμε τον τομέα αυτό της ε, βιοεισορροπίας από την υπολογισμό. Λοιπόν, είναι πολιτική λοιπόν η έκθεση. Δεν ε, βασίζεται ουσιαστικά σε πραγματική έκθεση του Αρεκτικού συνεδρίου. Και γι' αυτό δεν την αποδέχομαι και θα στείλω και στην διάσκεψη των Προέδρων μια επιστολή. Αυτό που μου λείπει είναι η επικέντρωση στην οικονομία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα εισοδήματα των ε, γεωργών και αυτό δεν το βλέπω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, βλέπω πολλά άλλα ζητήματα που αναφέρονται. Το πιο σημαντικό όμως της επιβίωσης των γεωργών είναι εντελώς παραμελημένο. Και Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Κρυντόρφμαν στη συνέχεια του έργου του, ε, γιατί έχει ακούσει πάρα πολλέ παρατηρήσει. Πώ θα τα συνενώσει όλα αυτά, δεν ξέρω. Καλή επιτυχία του, εύχομαι. Να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε ο καθένα λίγο στο θέμα του. Άκουσα και ανακοινώσει τύπου από την πατρίδα μου και άλλου που κάνουν διαφορετικά έργα εκτελούν από πολιτικές απόψεις. 30 Μαρτίου του επόμενου έτους. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και με τη μεταβατική φάση. Να σας, εξασφαλ... σας διαβεβαιώσω όμως ότι μέχρι τότε θα εργαστώ επικοδομητικά. Και η Πρωθυπουργό ε, με χθες, ε, ανάξω ότι είπε ψάχνει και θέλει πιο πολύ μεταβατική περίοδο και όχι λιγότερη. Δεν ξέρουμε φυσικά τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ακούω όλο και πιο πολλά για την γραφειοκρατία και για την απλοποίηση που χρειάζεται. Όλο αυτό λένε. Πώ θα τα βελτιώσετε λοιπόν αυτά. κανεί δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Είναι το ίδιο πρόβλημα έχουμε και με του γεωργού. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευρώπη είναι καλό. Να υπάρχει διαφορετική σχέση μεταξύ των Βρυξελών και των κρατών μελών και των περιφερειών. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις σχετικές πολιτικές είναι οι διαφορετικές ερμηνείες που δίνουν τα διαφορετικά κράτη-μέλη και μάλιστα και στο εσωτερικό των κρατών μελών πολλές φορές οι περιφερειές ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο και υλοποιούν με διαφορετικό τρόπο τις πολιτικές και όλοι φοβούνται, φοβούνται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κατηγορίες για απάτη, και τις κυρώσεις. Λίγες είναι οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη που σε κάποια που δεν έχουν ε, κυρώσεις κάθε χρόνο. Όχι επειδή είχαν σκοπό να προκαλέσουν προβλήματα, αλλά επειδή η υλοποίηση και η εφαρμογή δεν ήταν 100% κατά τη στοιχεία αυτών που θα επιθυμούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρόεδρε, θα ένα πάρα πολύ επίκαιρο και επίμαχο ζήτημα χτε. Γιατί όλο και πιο λίγοι είναι οι νέοι που στρέφονται και ασχολούνται με τη γεωργία. Εγώ δεν θα είμαι εδώ σε πέντε χρόνια, αλλά θα είναι εδώ στο Κοινοβούλιο οι βουλευτές θα ασχολούνται με το θέμα αυτό σε 5-10 χρόνια και ξανά και ξανά. Είναι απλό. Γιατί να γίνει κανείς γεωργός όταν είναι νέος, όταν βλέπει τους φίλους του που τελειώνουν το σχολείο να έχουν και καλύτερη ζωή και καλύτερη δουλειά, να μην δουλεύουν 7 μέρες ε, την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, όλες τις ε, αργίες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ φοβάμαι ότι αν θέλουμε να ε, σπρώξουμε τους, νέου νέους στη γεωργία, χρειάζεται μεθάρρυνση. Και ένα πράγμα ενθαρρύνει τον κόσμο να εργαστεί πιο πολύ και πιο σκληρά από τους άλλους είναι το χρήμα, το κέρδος. Όσο του λοιπόν ε, τα έσοδα είναι σωστά, όταν μιλάμε για κάποιον, γιατί δεν τον, ε, το, το, γιατί περνάμε σε τελική ανάλυση. Γιατί πολλοί, σε πολλούς δεν αρέσει. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται να αρέσει σε όλους. Και μπορεί κάποιοι να διαιρέσουν τα βαρτεμάχια τους και να θεωρηθούν δύο επιχειρήσεις, τι να του πω, καλή επιτυχία άμα το θέλουν να το κάνουν αυτό. Πολύ απλά κάποιοι παίρνουν παραπάνω από ό,τι άλλοι και αυτό θα πρέπει να σταματήσει γιατί δεν δίνει κίνητρα στους νέους και δεν επενδύει στο μέλλον. Ο μοναδικός τρόπος για να επενδύσουν οι νέοι Πώς θα το κάνουν αν δεν έχουν χρήματα. Θα πρέπει να πάνε σε μία τράπεζα, να ε, ε, καταθέσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να εργαστούν σκληρά για να το υλοποιήσουν στην επόμενη 20 αιτια 30 αιτία. Αυτή είναι η πρόκληση που έχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχουμε και εμείς, που έχουν και τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες. Γιατί όλοι είμαστε μαζί στο ίδιο στην ίδια κατάσταση και θα πρέπει όλοι να ωφεληθούμε τελικά. Σας ευχαριστώ. Τώρα η νέα μας αντιπρόεδρος, η κυρία Ζωάνα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρο, Σίγουρα γινόμαστε μάρτυρες πολλών αλλαγών στη Γεωργία και λόγω μακροοικονομικών αλλά και γεωπολιτικών τάσεων που περιορίζουν ε, την ε, βεβαιότητα και την ασφάλεια στην αγορά. Και οι μεγάλες δοκιμάσεις τιμών στα γεωργικά προϊόντα είναι ανησυχητικέ. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει για να διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε και μια εύρυθμα λειτουργούσα γεωργία. Η Ρουμανία έχει από τις μεγαλύτερες γεωργικές εκτάσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγικότητά μας όμως είναι αρκετά χαμηλή, γιατί όλο και περισσότεροι ασχολούνται με τη γεωργία. Γι' αυτό και η γεωργία στη Ρουμανία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα ε, ε, σε ό,τι αφορά τις μεγάλες αλυσίδες που διακινούν μικρό τμήμα ρουμανικών προϊόντων λόγω του χαμηλού περιθωρίου κέρδους. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε την ανταγωνιστικότητα των Ρουμάνων Γεωργών στην ευρωπαϊκή αγορά. Εγώ είμαι υπέρ της διατήρησης του γεωργικού προϋπολογισμού και στους δύο πυλώνες και είμαι κατά των οροφών των ανωτάτων όριων. Επίσης, θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις άμεσες ενισχύσεις χωρίς εθνική χρηματοδότηση για να στηρίξουμε το γεωργικό εισόδημα. Και μέτρα όπως τα ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις και τη χρηματοδότηση από τον εθνικό προϋπολογισμό θα περιορίσουν την ικανότητα της κοινής γεωργικής πολιτικής να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια και στην εσωτερική αγορά. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποβάλλοντας και εγώ μία ερώτηση που άκουσα από τους Γεωργούς, ερώτηση, παρατήρηση, όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι εστί ε, στρατηγικό σχέδιο και το νέο τρόπο εφαρμογής, μας ακούν οι αγρότες ε, και λένε «εντάξει, έχουμε ε, το 30% του πρασινίσματος, ε, ε, βάλτε το στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο, αλλά το 70% μη μας το πειράζετε, γιατί αν πάρετε το 30% για το πρασίνισμα, αφήστε μας τουλάχιστον άθικτο το 70%. Αυτή είναι η ανησυχία των αγροτών μας. Αυτό τους ενδιαφέρει και αυτή, εκεί έγκυται η δυσαρέσκειά τους κατά κάποιο τρόπο με με τις προτάσεις. Πολύ πλούσια συζήτηση, πληθώρα ερωτήσεων κύριε Διευθυντά. Έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσους συνεισέφεραν στη συζήτηση. Εντυπωσιάστηκα στο τέλος με αυτά που είπε ο κ. Νίκολσον. Μου μίλησε αυτό που είπε έθεσε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Ανέφερα ανησυχίε που έχει γενική μου διεύθυνση και είχε γενική μου διεύθυνση όταν επεξεργαστήκαμε ε, το κείμενο της ανακοινώσεως. Να διατρέξω τις ερωτήσεις. Επικεντρωνόμενος επί των επαναληφθέντων θεμάτων. Αλλιώς θα κουβεντιάζουμε δυόμιση ώρες και δεν έχουμε χρόνο. Όσον αφορά το μοντέλο επίτευξη των στόχων και τα σχέδια ΚΑΠ, αρκετοί ομιλητέ αναφέρθηκαν στη σχέση μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών και ομοσπόνδων ε, κρατηδίων. κάτι κράτη-μέλη τα οποία είναι οργανωμένα περιφερειακά, σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι σαφές ότι οι συνταγματικέ απαιτήσει που απορρέουν από την όλη κατάσταση πρέπει να γίνουν σεβαστές. Γι' αυτό, με κάποιο τρόπο πρέπει να εξευρεθεί η δομή, η κατάλληλη για τα στατικικά σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη αυτές οι ιδιαιτερότητες. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται επεξεργασία και να αναφέρετε σαφώς την πρόταση που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι αυτό έχει σημειωθεί δεόντως όχι μόνο από τη συζητήσεις εδώ αλλά και από τη συζητήσεις στο Συμβούλιο. Είναι σαφές ότι πρέπει να φτιάξουν το κατάλληλο πλαίσιο ούτω ώστε να έχουν περιθώρια λιγμών οι περιφέρειες. Αυτό είναι σαφέστατο. Θα σταματήσω εδώ πάνω σε αυτό. Αν προχωρήσω περαιτέρω θα εκφράζω προσωπικές απόψεις. Αλλά οι προσωπικές μου απόψεις δεν αφορούν την παρούσα συζήτηση τέθη το εξή ερώτημα. Ποιο καθορίζει ποιο είναι ο δικαιούχο. Αυτό σχετίζεται με τη συζήτηση την παρελθούσα επί ενεργού ε, Γεωργού. Τώρα αποκαλείται πραγματικός γεωργό, γνήσιος γεωργό στην κοινούση. Επί σειρά ετών ε, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία. Εδώ, στο Κοινοβούλιο. Αλλά εκφράζεται και στην κοινωνία των πολιτών αυτή η ανησυχία. Αυτή η αφορά το εξή. Η γεωγραφική στήριξη χορηγείται στους δικαιούχους εκείνους που κανονικά δεν θα έπρεπε να παραλάβουν αυτή την ενίσχυση και πολύ δύσκολο να εντοπιστούν οι λόγοι για τους οποίους δεν έπρεπε να δοθεί στήριξη. Το 2013 στη μεταρρύθμιση που κάναμε καταρρίξαμε σε έναν κανόνα. Σύμφωνα με αυτόν εξαιρούνται δικαιούχοι που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ενεργοί ε, γεωργοί και έπρεπε να μπουν σε έναν αρνητικό κατάλογο. Προφανέστατα, στα πλαίσια του κανονισμού Omnibus αυτό καλύπτεται. Ήταν γραφειοκρατικό το όλο πρόγραμμα το πλαίσιο, γραφειοκρατικοί κανόνες που καμιά φορά έπληταν και τους αθώους. Και γι' αυτό εφαρμόζεται προαιρετικά. Και τα κράτη-μέλη έτσι έχουν τη δυνατότητα, όταν θεωρούν ότι υπάρχει πραγματική επιτόπια ανάγκη, να χρησιμοποιούν το κατάλληλο μέσο. Εν τω μεταξύ, έχουν τεθεί και άλλα σημεία. Φερρυπίν, οι επενδυτές που γίνονται μεγάλοι γεωκτήμονες, είναι ιδιοκτήτες μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Άρα η ζωή κεφαλαίων που δεν προέρχονται από τη Γεωργία, δεν σχετίζονται με τη Γεωργία μέσα. Αυτό είναι μια ακόμη ανησυχία. Άρα και αυτό μπορεί να ενταχθεί στην όλη έννοια του πραγματικού, του γνήσιου γεωργού. Πολύ δύσκολο αυτό ο όρο να γίνει επιχειρησιακό όρο και να εισαχθεί σε νομοθεσία. Εργαζόμαστε σκληρά επ' αυτού. Να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί. Εν πάση περιπτώσει, στο μοντέλο αυτό επιτεύσεω στόχων, τα κράτη-μέλη θα έχουν μεγαλύτερη επικουρικότητα. Θα μπορούν να καθορίσουν τι αποτελεί γνήσιο Γεωργό και θα ήταν λογικό. Τι είδαμε στο παρελθόν ότι έχουμε διαφορετικές καταστάσεις διάφορα κράτη-μέλη και τα προβλήματα των κρατών μελών ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Σε μια χώρα ίσως το πρόβλημα να είναι επενδύσεις. Σε άλλη χώρα ότι είναι περιθωριακή επιχείρηση η γεωργία, δεν είναι στο επίκεντρο του επιχειρηματικού κόσμου. Χρειάζεται μεγαλύτερη επιχειρη... ε, συγγνώμη, επικουρικότητα για τα κράτη-μέλη, να μπορούν καθώς τα κράτη-μέλη τι εννοεί αυτός ο όρος. Και αυτή είναι η λογική που ακολουθήθηκε και στη διαδικασία Omnibus. Άλλη ερώτηση. Δείκτες. Αν θα εισαχθούν νέοι δείκτες τώρα. Ε, δείκτες αντικτύπου ή δείκτες αποτελεσμάτων και υπονοήθηκε ότι τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Που σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει πραγματιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τέτοια δήλωση. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε δημιουργήσει συστήματα επιδόσεων για το δεύτερο πυλώνα, πολύ πιο προθυμένα συστήματα από ό,τι στον πρώτο πυλώνα. Το 2013 στη μεταρρύθμιση που κάναμε, Δημιουργήθηκε κοινό πλαίσιο για αξιολόγηση και παρακολούθηση. Εκεί περιέχονται πολλοί δείκτες, πολλών τύπων και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της πολιτικής. Ποιο είναι το προβλήμα των δικτών, ότι είναι πολυάριθμοι. Και θα προσπαθήσουμε στην όλη διαδικασία να μειώσουμε τον αριθμό των δικτών και να επιλέξουμε τους ρεαλιστικότερους και βέλτιστους, προσπαθώντας πάντο να μην επανεφευρίσκουμε δείκτες για τους οποίους δεν θα διαθέτουμε πηγές στοιχείων, διότι τους δείκτες που έχουμε έχουμε στοιχεία. Αυτή ε, είναι συνεχιζόμενη εργασία και έχουμε προδέψει πάνω σε αυτό. Θέλουμε να έχουμε έναν κατάλογο δικτών. Ο κατάλογος θα είναι περιορισμένος σε αριθμό δικτών θα βασιζόμαστε στους υφιστάμενους πόρους πληροφοριών και στοιχείων. Και έτσι οι δείκτες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η ε, κυρία Ροδρίγκες επέκρινε την ΚΑΠ απευθυνόμενη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ να πω κάτι απλό. Η μεταρρύθμιση του 2013 αποτελεί την βάση της τρέχουσης ε, πολιτικής που διαχειριζόμαστε μαζί με τα κράτη-μέλη. Υιοθετήθηκε από τον νομοθέτη και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο με μεγάλες πλειοψηφίες. Νομίζω ότι όλοι είμαστε στην ίδια βάρκα. Εάν ε, θέλουμε να βελτιώσουμε την όλη κατάσταση αν κρίνουμε ότι δεν είναι καλή. Μία από τις πτυχές που αναφέρθηκε ήταν ανανέωση γενεαλογική. Η Νέη Γεωργία, ο κ. Νίκολσον ανέφερε πολλά καλά στοιχεία πάνω σε αυτό. Η ανανέωση αυτή των γεωργών, η γενεαλογική, αντιμετωπίζει στην ανακοίνωση το κατέστησε ηλίου φαϊνότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη σημαντική πτυχή για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Πώς οι νέοι γεωργοί οι νέοι να αποφασίσουν να γίνουν γεωργοί. Όπως είπε ο ο Νίκολσον, γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα που δεν θέλουν οι νέοι να γίνονται γεωργοί. Τα αίτια ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Μου λένε από διάφορες χώρες ότι ο βαθμός δυσκολίας όσον αφορά τους νέους που γίνονται γεωργοί ποικίλει. Υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη όπου οι νέοι ε, γίνονται γεωργοί. Σε άλλες χώρες τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ε, επί τη βάση ενός ρεαλιστικού ευρωπαϊκού πλαισίου θα ήταν καλό τα κράτη-μέλη να μην εφαρμόζουν μια γενική πολιτική, αλλά να αντιστοιχούν τις προσπάθειες που καταβάλουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται όσον αφορά την ε, απασχόληση των νέων στον γεωρικό τομέα. Αναφέρεται ότι η ανακοίνωση δεν ε, περιέχει αρκετά στοιχεία για την κατάσταση στις αγορές και ότι δεν ε, αποτελεί σε επαρκή βαθμό οικονομική πολιτική. Να απαντήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκαθαρίσει και έχει βάλει την ε, θέση του Γεωργού στην αλυσίδα τροφίμων ε, στην ατζέντα τη, σε μεγάλο βαθμό μάλιστα. Ήμασταν όσο πιο γρήγοροι μπορούσαμε σε ό,τι αφορά τη σχετική νομοθεσία, σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της θέση ε, των τετάξεων ανταγωνισμού στην ΚΟΑ. Πλέον αυτό περιλαμβάνεται. Το πακέτο για το γάλα το έχει ήδη κάνει αυτό το 2011 για την αγορά γάλακτος. Χρησιμοποιείται, αλλά όχι επαρκώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή τη ε, μιλάει για μια πιο επικεντρωμένη υποστήριξη εισοδήματο που ακριβώς ως σκοπό έχει να βελτιώσει την κατάσταση όσων χρειάζονται πιο πολύ στο πλαίσιο της ε, ΚΑΠ, συστήματα αναδιανομής των πληρωμών όπως ε, υπάρχουν ήδη και αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση. Αυτό αποτελεί μία πτυχή μόνο το θέμα του γνήσιου γεωργού. Επίσης παίζει το ρόλο του και γενικά όσο πιο επικεντρωμένη, όσο πιο στόχοθετημένη γίνεται χρήση των συστημάτων ενίσχυσης. Αυτό κινείται προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να εξουδετερώσει την ανάγκη για τα όσα θα πρέπει να προβάλλουμε. Και ήταν αποφασίζει και η πολιτική των ε, νομοθετών ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι μια πολιτική η οποία προσανατολίζεται στην αγορά. Θέλει ο γεωργός ε, στην ευρωπαϊκή αγορά να είναι ανταγωνιστική. Αυτό επικρίνεται σε κάποιες περιπτώσεις, όπως και σήμερα, παρελπτόντως στη συζήτηση, ότι είναι μια πολιτική που προσανατολίζεται και στην εξαγωγή προϊόντων. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι καθαρή η ισορροπία σε ό,τι αφορά εισαγωγών και εξαγωγέ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια αρκετά σημαντικά. Ο προσανατολισμό στι εξαγωγέ είναι κάτι το οποίο δημιουργεί αξία στην εσωτερική αγορά. Είναι κάτι που δίνει επιπλέον ε, αγορές ε, για τα προϊόντα που παράγονται στην ε, Ευρώπη. Εντάλλως, ε, αν δεν υπήρχε αυτή η διάσταση, θα συρρυκνωνόταν η γεωργική αγορά και θα μειωνόταν η δυνατότητα δημιουργίας ε, προστιθέμενης αξία ε, στον κλάδο. Αυτό είναι μία από τι βασικές θέσεις της ΚΑΠ που ακολουθείται επί σειρά ετών, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Και γι' αυτό λοιπόν αποτελεί ακρογωνία λίθο της ανακοίνωση. Θα πρέπει να υπάρχει φυσικά καλύτερη στόχευση, επαναλαμβάνουμε, τη ενίσχυση και θα πρέπει να φροντίσουμε καλύτερα κάποιους παραγοντές. Αναφέρθηκε στη συζήτηση αυτή επίσης από κάποιους ομιλητές ότι η τρέχουσα ΚΑΠ δεν αποτελεί μοντέλο και υπόδειγμα ομοιογένειας. Εμείς σε διάφορες περιστάσεις ξεκαθαρίσαμε ότι κοιτώντας τον πρώτο πυλώνα έχουμε 60-70 διαφορετικές ε, εναλλακτικές από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν τα κράτη-μέλη. Έχουμε σε ό,τι αφορά την εθελούσια υποστήριξη πάνω από 200 διαφορετικά συστήματα ενισχύσεων που έχουν εφαρμοστεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση, όπως αναφέρθηκε για παράδειγμα, από διάφορους ομιλητές, αυτό οδηγεί, επαναλαμβάνω, σε μια κατάσταση όπου υπάρχει ήδη πραγματική πιθανότητα στρέβλωσης της αγοράς. Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει ένα σύστημα χωρίς εθελούσια υποστήριξη και το διπλανό κράτος μέλος εξαντλεί τα ανώτατα όρια σε ό,τι αφορά την υποστήριξη αυτή, προφανώς στις συνοριακές περιοχές θα ανακύψουν προβλήματα, ενδεχομένως σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα των μεν έναντι των δε. Περιγράφεται το status quo, την κατάσταση, όσο έχει τώρα. Όχι στο μέλλον. Ήδη, από τώρα. Νομίζω ότι είναι όνειρο αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών που θέλει να δώσει ευελεξία στα κράτη-μέλη, αλλά είναι όνειρο πατέρα να πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε κάποιες περιπτώσεις, σε καταστάσεις που θα αγγίζουν τα όρια της τρέβλωσης. Και σε ό,τι αφορά το μοντέλο απόδοσης, ε, το delivery model. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήδη υπάρχει και δεν θα αμα, ε, υποχωρήσει. Δεν θα μπορέσουμε να κινηθούμε προς το μοντέλο της λιγότερης επικουρικότητα, της λιγότερης ευελιξίας. Δεν είναι δυνατόν. Και αναφέρθηκε ότι το ευημερία των ζώων δεν τονίστηκε επαρκώς. Εγώ το ανέφερα σήμερα στην παρουσίασή μου και νομίζω ότι αναφέρεται και στην ανακοίνωση. Και ασφαλώς η ευημερία των ζώων ήδη αποτελεί τμήμα της πολλαπλής συμμόρφωσης και τετάξεις για την ευημερία των ζώων συμπεριλαμβάνονται στην πολλαπλή συμμόρφωση. Αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες και οι εκτροφείς που δεν σέβονται αυτά τα κριτήρια δεν λαμβάνουν πλήρη υποστήριξη. Τώρα, η ουσιαστική νομοθεσία για την ευημερία των ζώων είναι εκτός του πλαισίου της ΚΑΠ. Αυτό το αντιμετωπίζει η DG Sante, η Γενική Διάθεση Sante και αυτό νομίζω ότι θα ήταν το πρώτο σημείο εκκίνησης αν θέλετε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της ΚΑΠ. Ουσιαστικά να προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε τους υφιστάμενους κανόνες μέσω, για παράδειγμα, της πολλαπλής συμμόρφωσης, προκειμένου να είναι πιο απλή η συμμόρφωση και να προσφέρουμε συστήματα ενίσχυσης, ιδιαίτερα στον δεύτερο πυλώνα, όπου τα κρατημέλη είναι σε θέση να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν μέτρα φιλικά προς την ευημερία των ζώων, τα οποία θα υπερβαίνουν την προβλεπόμενη νομοθεσία. Και αυτό ακριβώς έχει ο σκοπό και θα έπρεπε να έχει ο σκοπό και στο μέλλον η πολιτική. Άρα, δεν το απορρίπτει αυτό η ανακοίνωση ή οι ιδέες που έχει εκφράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελλοντική ΚΑΠΑ. Κύριε Χόισλινγκ, είπατε ότι έχετε την εντύπωση ότι η ανακοίνωσή μας βασίζεται το ότι δεν τα καταφέρουμε εμεί από μόνοι μα, γι' αυτό τα σπρώχνουμε όλα στα κράτη-μέλη. Ο κύριο Νταντάν είπε επίση ότι ουσιαστικά η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην DG Agri ε, έχει λιγότερο προσωπικό και δεν θέλει να κάνει τη δουλειά της. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν είναι ότι δεν τα βγάζει πέρα. Πολύ απλά, οι πολιτικές τα τελευταία χρόνια έχουν επικριθεί όλο και πιο πολύ ότι είναι περίπλοκες και εκ παραλίλου, επίσης έχει ασκηθεί έντονη κριτική κατά της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Επιτόπου σε ό,τι αφορά τις κυριώσεις, σε ό,τι αφορά τις ε, διορθώσεις, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ε, δεν έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα ζητήματα πολιτικής, αλλά με υλοποίηση, ακόμα και τεχνικών κανόνων σε κάποιες περιπτώσεις. Το ερώτημα λοιπόν που θα πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας δεν είναι κατά να έχει μειωθεί το προσωπικό μας και έχουμε επιβαρυνθεί υπερβολικά. Και να σας ε, ε, διαβεβαιώσω ότι το delivery model θα μας απασχολήσει επισταμένως, θα μας επιβαρύνει πολύ. Το θέμα είναι κατά πόσον μπορούμε να βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή ε, μεταξύ του τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το τι θα γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι σημαντικό ζήτημα και το είπατε και εσείς κύριε Χόισλινγκ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι 80% της ε, περιοχής καλύπτεται από το πράσινο προσανατολισμό και ότι το ελεκτικό συνέδριο είπε 5% μόνο. Δεν είπε αυτό το ελεκτικό συνέδριο, είπε ότι 5% των εκτάσεων σημειώνουν ε, πρόοδο. Μία προσπάθεια παραπάνω από όσα συνέβαιναν έω τώρα. Αυτό ήταν το συμπέρασμα και το πόρισμα του ελεκτικού συνεδρίου. Σωστό, η λάθο είναι άλλο θέμα. Δεν μίλησε όμω για το τι ποσοστό της έκτασης καλύπτεται από το πρασινισμά. 80% καλύπτεται. Όντως, το θέμα είναι που επιτέχθηκε ο σκοπός της πράσινης ε, προσέγγισης. Επίσης, το ελεγκτικό συνεδρίο είπε και κάτι άλλο, το οποίο δεν το αναφέρεται, το οποίο είναι ότι το η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό ήταν πολύ πιο φιλόδοξη σε σχέση με το προτινόμενη νομοθεσία. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί υποδεικνύει ένα βασικό πρόβλημα στον κλάδο. Ότι μια πρόταση η οποία ήταν μάλλον άμεση και απλή αποδυναμώθηκε με ένα σωρό εξαιρέσει και εναλλακτικέ λύσει. Και τώρα έρχεται να μας βάλει βαθμούς στο ελεκτικό συνέδριο δεν ξέρω τώρα αν είναι πολιτικά τα κίνητρα του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά τα πορίσματα τα οποία βλέπουμε είναι σαφή. Στην ανακοίνωση λοιπόν και γι' αυτό δίνεται έμφαση ιδιαίτερος στους περιβαλλοντικού ε, στόχους. Αν... Αναφέρεται ότι θα θέλαμε να απομακρυνθούμε από ένα σύστημα που κατά τη γνώμη πολλών δεν ε, υλοποίησε τους στόχους του και τα αναμενόμενα και να το απλουστεύσουμε πρώτα και να, το, και να ενσωματώσουμε τα βασικά κριτήρια και τις βασικές προϋποθέσεις για τον οικολογικό προσανατολισμό, κάπως πιο ενισχυμένους, με μεγαλύτερες φιλοδοξίες ε, και αιρεσιμότητα και να το χρησιμοποιήσουμε ως βασικό σενάριο για τον δεύτερο πυλώνα. Και αυτό είναι απλούστερο, μια και η πολλαπλή συμμόρφωση είναι αρκετά αποτελεσματικό σύστημα και ίσως υπόσχεται πολύ περισσότερα ε, και έχει πολύ περισσότερο δυναμικό από το ισχύον. Αναφέρθηκε, κύριε Δεκάστρο, από εσάς αν δεν κάνω λάθος, ε, μήπως το στρατηγικό σχέδιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγχρηματοδότηση στον πρώτο πυλώνα. Νομίζω ότι η συγχρηματοδότηση του πρώτου πυλώνα είναι ένα θέμα που θα εξαρτηθεί από τη λύση που θα δοθεί στο ΠΔΠ, στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν αναφέρεται στην τελευταία ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και ίσως είναι αυτό μια καλή ένδειξη. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με το κατά πόσο θα έχουμε στρατηγικό σχέδιο και το πώς θα διαρθρωθεί αυτό. είναι κάτι που δεν είναι ρεαλιστικό. Ο κύριος Κολομπιέ, αν λέω σωστά το όνομά του, υπενήχθηκε ότι η πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να καταργήσει τις άμεσες ενισχύσεις. Όχι, καθόλου. Φαίνεται ακριβώς από την ανακοίνωση ότι δεν είναι καθόλου αυτή η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ε, Επιτρόπου, γιατί θεωρούμε τις άμεσες ενισχύσεις στον ακρογωνιαίο λίθο της στήριξης ε, ε, εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να διαδραματίζουν και στο μέλλον αυτό το ρόλο οι άμεσες ενισχύσεις. Απλώς θέλουμε ένα πιο στοχευμένο σύστημα που θα προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες των αγροτών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους και τις ε, διαφορετικές καταστάσεις των περιφερειών και των κρατών τους. Ο ρόλος του νομοθέτη στη διαδικασία αυτή θα είναι ο ίδιος όπως και στο παρελθόν. Δηλαδή θα πρέπει ο νομοθέτης να ε, διαδραματίσει το έπακρο το ρόλο του, να αποφασίσει δηλαδή για, τους, ε, για τις βασικές νομοθετικές πράξεις με το περιεχόμενό τους, είτε κατά παραδοσιακό τρόπο μέχρι το, όπως αυτό που υιοθετήσαμε το 2013 είτε με το νέο delivery model που περιλαμβάνει η ανακοίνωσή μας. Ο νομοθέτης θα αποφασίσει αν η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επιθυμητή και πώς μπορεί να αποτυπωθεί σε νομικό κείμενο. Δεν βλέπω καμία διαφορά σχέση με το παρελθόν. Ο νομοθέτης και πάλι θα έχει το τελευταίο λόγο για τα θέματα αυτά. Και εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία και την περαιτέρω συζήτηση. Αναφέρθηκαν ε, ζητήματα όπως η σύγκληση, εξωτερική σύγκληση. Δεν θα τα σχολιάσω, γιατί συνδέονται εγγενώς με τη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και σίγουρα σε αυτό το πλαίσιο θα επαναφανιστούν και πολύ πιο διεξοδικά και έντονα. Ο κύριος Λίντς έθεσε τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορούσε τα χαρακτηριστικά, την αρχιτεκτονική του σχεδίου της ΚΑΠ. Βέβαια, η θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι συνταγματικές διατάξεις των κρατών μελών, εννοείται. Κάτι που ε, προϋποθέτει τη συμπερίληψη του περιφερειακού ή του ομοσπονδιακού επίπεδου στη Γερμανία ή των περιφερειών σε άλλες χώρες. Τη συμπερίληψη αυτό λοιπόν με τον κατάλληλο τρόπο στο εθνικό σχέδιο. Δεν μπορώ να σας πω εγώ ξεκάθαρα πώς θα συμβεί αυτό. Πάντως σίγουρα αυτό μας ενδιαφέρει και ε, έχουμε επίγνωση ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, ε, θεωρούμε και γνωρίζουμε ότι αυτή, αυτή η πρόταση σε καμία περίπτωση θα πρέπει να καθυστερήσει τη διαδικασία. Δηλαδή να μην περιμένουν όλοι τον πιο αργό κρίκο της αλυσίδας και της διαδικασίας. Αλλά θα πρέπει να διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να είναι λειτουργικός και να μην παρεμποδίζει την πρόοδο. Ο κύριος Λίνς ρώτησε αν όντως το greening μπαίνει στο δεύτερο πυλώνα. Η απάντηση είναι όχι. Η ιδέα δεν είναι να μπει το greening στο δεύτερο πυλώνα, αλλά να συμπεριληφθεί σε ένα βασικό επίπεδο αιρεσιμότητας που θα ακολουθεί την λογική της πολλαπλής συμμόρφωσης του παρόντος κανονισμού της παρούσας Επίσης ρωτήσατε αν ο, δεύτερος, πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας θα συνδυαστούν, θα γίνουν verknüpft, όπως λέμε στα γερμανικά, αν είναι αλληλένδετοι. Μα είναι ήδη αλληλένδετοι οι δύο πυλώνες. Γιατί η ΚΑΠ είναι ενιαία πολιτική που απαρτίζεται από δύο πυλώνες, τον πρώτο και τον δεύτερο. Πάντως, στο μέτρο του δυνατού θα συνδεθούν και με ένα στρατηγικό σχέδιο και από το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της διαδικασίας προγραμματισμού θα θεσπίσουν στόχους που θα τους υλοποιούν με μέτρα είτε του πρώτου είτε του δεύτερου πυλώνα. Και υπάρχει και το οικολογικό, οικοπεριβαλλοντικό περιβαλλοντικό στοιχείο. Εκεί τα κράτη-μέλη θα αποφασίζουν αν θέλουν ένα ενδιάμεσο οικοπεριβαλλοντικό στοιχείο, ένα σχέδιο για τα θρεπτικά συστατικά, ε, και ο θελός όμως τον πρώτο πυλώνα. Και θα μπορούν επίσης για τα σχέδια για τα θρεπτικά συστατικά να τα, ε, να τα συμπεριλαμβάνουν στο δεύτερο πυλώνα. Αυτό όμως το αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Δική τους είναι η επιλογή και η ευχέρεια και αυτό έχει νόημα και στα πλαίσια της επικουρικότητας. Η κυρία Μαγκίνες ε, ρώτησε ποιο είναι το βασικό σενάριο. Το βασικό σενάριο είναι κυρίως η αιρεσιμότητα. Αυτό είναι το πρώτο στρώμα, το πρώτο επίπεδο. Θυμάστε και τον πίνακα. Φυσικά θα πρέπει να γίνεται σεβαστό το βασικό σενάριο και να το ξεπερνάμε και όλα. Επίσης, ρωτήσατε αν οι άμεσες ενισχύσει ε, θα δίνονται με βάση τη γη. Τίποτα στην ανακοίνωση δεν εμποδίζει κάτι τέτοιο στο μέλλον ή δεν υπονοεί ότι δεν θα ισχύσει αυτό στο μέλλον. Ούτε ότι δεν μπορεί να υπάρχει κατα, καταποκοπή ενίσχυση ένα εκτάριο. Πάντως όλες οι πληρωμές θα σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις σε δυνάμει της αιρεσιμότητας. Είπατε ότι δεν θα πρέπει να πληρώνουμε για νέους οικοτόπους, αλλά για τους ε, υφιστάμενους οικοτόπους. Και εδώ επανέρχομαι στο σχόλιο του ελεκτικού συνεδρίου, το ανέφερα και προηγουμένως, απαντώντας τον κύριο Χόισλινγκ. Το θέμα είναι, η αύξηση της περιβαλλοντικής μας φιλοδοξίας σημαίνει ότι ξεπερνάμε τις ισχύουσες διατάξεις και ε, ε, αυξάνουμε το περιβαλλοντικό πλεονέκτημα της ΚΑΠ από ό,τι ισχύει μέχρι τώρα. Τι να σας πω, εγώ δεν έχω ε, ορισμό για το τι εστί δίκαιη μεταχείριση. Αυτή είναι μάλλον πολιτική συζήτηση που θα γίνει μεταξύ των νομοθετών βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως γνωρίζω ότι στη δημόσια συζήτηση αλλά και στην πολιτική συζήτηση η ιδέα μιας δίκαιης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων ε, ανακύπτει συχνά. Και το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το σχέδιο ψηφίσματος για την απαλλαγή. Εκεί ε, καλείται έντονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τη δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων στις προτάσεις της. Και αυτή η δικαιότερη κατανομή συνδέεται πολύ συχνά με το παράδειγμα του 80-20. 80%, 80 των αγροτών λαμβάνουν το 20% των ενισχύσεων. Βέβαια, η κατανομή των αγροτεμαχίων και αυτή παρακολουθεί το λόγο 80 προς 20, δηλαδή 20% των αγροτών ε, κατέχουν το 80% της γεωργικής γης. Οπότε, απριόρι, σε ένα σύστημα που συνδέεται με τη γη, είναι λογικό ότι 80% των ε, ενισχύσεων πάει σε 20% των γεωργών, μια και έχουν το περισσότερο ποσοστό της γης. Αλλά 71% της ενίσχυσης πηγαίνει σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν 5 με 250 εκτάρια. Οπότε αλλάζει η αντίληψη εδώ με αυτό το στοιχείο, γιατί σχεδόν το σύνολο, το 80% των ενισχύσεων πηγαίνουν σε ε, εκμεταλλεύσεις που είναι μικρές, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, φυσιολογικές, με διάφορα βέβαια μεγέθη, διάφορες διαστάσεις, γιατί σε μερικές περιπτώσεις, σε μερικές χώρες οι γεωρικέ εκμεταλλεύσεις είναι πιο μικρές, ενώ σε άλλες είναι πιο μεγάλες. Σε πολλά μέρη της Γερμανίας ε, ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις 100-150 εκταρίων θεωρούνται φυσιολογικές, συνηθισμένες. Οπότε δεν θα πρέπει να αντλούμε βιαστικά συμπεράσματα από αυτό το λόγο 80 προς 20, αλλά να τα εξετάζουμε ευρυθέστερα. Πάντως, σίγουρα θα πρέπει να δούμε τους μεγάλους δικαιούχους που λαμβάνουν εκατομμύρια ευρώ από την ΚΑΠ και να διαρωτηθούμε, το κάνουμε και στις προηγούμενες προτάσεις, αν Υπάρχουν οικονομίες κλίμακος ε, που δικαιολογούν μία σταδιακή μείωση, προοδευτική μείωση ή θέσπιση ανώτατου ορίου, το κάπινγκ, θέσπιση κάποιων οροφών. Πλησιάζω σχεδόν προς το τέλος. Ε, μία πολύ σημαντική ερώτηση που τέθηκε είναι αυτή της μετάβασης. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ δύο καταστάσεων. μερικοί υπενήχθησαν ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι την εκλογή του νέου Κοινοβουλίου για τη διεκπαιρέωση των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Γιατί αυτή η περιπτώση θα συνεχιστούν και στο μέλλον οι διαπραγματεύσεις αν δεν ολοκληρωθούν σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Τώρα, πότε δεν ξέρω. Μέχρι πότε. Αν δεν είμαστε έτοιμοι εγκαίρως να εφαρμόσουμε την πολιτική από το 2021. Φυσικά θα χρειαστούν σε τέτοια περίπτωση κάποια μεταβατικά μέτρα. Το ίδιο είχαμε και στην προηγούμενη ε, μεταρρυθμίση. Και εκεί είχαμε μεταβατική νομοθεσία που την ενέκριναν οι νομοθέτες. Και αν διαπιστώσουμε τέτοια καθυστέρηση θα υποβάλουμε μεταβατικές προτάσεις. Αν όλα όμως πάνε ε, κατευχήν και με βάση το χρονοδιάγραμμα, πόσο χρόνο θα χρειαστεί για την εφαρμογή των αποφάσεων σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό το νέο μοντέλο, το νέο delivery model. Και εκεί θα χρειαστούμε ε, επαρκώς μακροχρόνια μεταβατική περίοδο, ώστε να μπορέσουν όλα τα επίπεδα να εφαρμόσουν αυτό το νέο πλαίσιο. Και άρα αρκετό χρόνο χρειάζονται και τα κράτη-μέλη και οι φορείς πληρωμών και οι εγρότες για να καταλάβουν τι τους γίνεται για να καταλάβουν ποια είναι η θέση τους στο όλο νέο σύστημα, αλλά χρειάζεται χρόνος και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το λέω με ταπεινοφροσύνη, γιατί παρόλο που δεν είμαστε εδώ στην πρώτη γραμμή της συζήτησης και εμείς θα πρέπει να δούμε ε, να βρούμε κάποια σημεία αναφορά και να δούμε πώ θα εγκριθούν τα εθνικά σχέδια. Δεν μπορούν αυτά να γίνουν μία ανοιχτή. Ελπίζω να κάλυψα τι περισσότερε ερωτήσει. Αν ξέχασα μερικέ, σα ζητώ συγγνώμη. Αλλά θα έχουμε και στο μέλλον ευκαιρίε για να επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κύριε Μέγκελε. Και με την υποβολή των ερωτήσεων θέλαμε ακριβώς να θίξουμε κάποια προβλήματα για να σας επιστήσουμε την προσοχή στα προβλήματα αυτά και να τα λάβετε υπόψη και στο μέλλον. Δεν θέλαμε να μας δώσετε απαντήσεις αμέσω. Δεν ήταν αυτός ο στόχος της συζήτησης, απλώς να επισημάνουμε τα προβλήματα για να τα λάβετε υπόψη. Γι' αυτό και ήταν τόσο πλούσια και ευρία η συζήτηση. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε. Πάντως και αν έχουμε και άλλες απορίες και άλλες ερωτήσεις θα τις ε, στείλουμε στους εμπειρογνώμονές μας, αλλά θα τις αποστείλουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντόρφμαν. Πάντως νομίζω ότι ήταν καλή και επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντόρφμαν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίσπευση των εργασιών, γιατί ε, εργαζόμαστε παράλληλα με ταχύς και αυτό περνίζεται θετικό μέλλον. Τώρα, και αν τα καταφέρουμε να τα διεκπαιρεώσουμε όλα πριν τι ευρωεκλογέ, θα έχουμε περισσότερο χρόνο για τις εργασίες ε, και τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών για την ε, ε, εκπόνηση των εθνικών στρατηγικών σχεδίων. Φυσικά δεν είναι και εύκολα αυτά, αλλά έτσι είναι η ζωή, δύσκολη ζωή. Εφτά, ευχαριστώ πάντως σε όλους για τη συζήτηση και δεν ξέρω αν ο κύριος Δόρφαν θέλει το λόγο για να κάνει μια σύντομη ανακεφαλαίωση και σύνοψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, και να κλείσω εν συντομία. Νομίζω ότι του περιεχομένου δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ εκτενής και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έγινε για το περιεχόμενο στις 12 Μαρτίου στο Στρασβούργο θα παρουσιάσω την έκθεση και τότε θα γίνει και πάλι μια συζήτηση επί του περιεχομένου της έκθεσης. Αυτό που ήθελα μόνο να κάνω είναι να παρακαλέσω τους συναδέλφους να διαβάσουν το σχέδιο της έκθεσης και να προσπαθήσουμε τις επόμενες εβδομάδες να εργαστούμε επικοδομητικά επί των τροπολογιών. Όπως σας είπα, εγώ ε, προφανώς είμαι στη διάθεσή σας και το γραφείο μου ολόκληρο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα προκειμένου στο τέλος του Μαΐου να έχουμε έτοιμη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό για τα βασικά ζητήματα τα οποία πολλοί ανέφεραν σήμερα να τοποθετηθεί με σαφήνεια το Κοινοβούλιο καθότι ως συνομοθέτης είμαστε υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και την υλοποίηση τέτοιων σημαντικών νομοθετικών προτάσεων. Να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω πολύ, να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απαντήσεις τους. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Ντόρφμαν και σας και τους συνεργάτες σας. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανα σκόπιμο να μην περιορίσω τη διάρκεια της συζήτησης, ώστε να μπορέσουμε όλοι να παρουσιάσουμε τα σχόλιά μας, ε, τις απόψεις μας και τις ερωτήσεις μας. Αλλά ο χρόνος περνά. Ας περάσουμε λοιπόν και εμείς ε, στο τελευταίο συστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, το υγεία είναι μία. Καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Ο συντάκτης γνωμοδότης είναι ο κύριος Κάρθη. Όπως ξέρετε αποφασίσαμε ε, να λάβουμε υπόψη το θέμα της μικροβιακής αντίστασης στα, στην κτηνοτροφία για να περιορίσουμε το, ε, το φαινόμενο αυτό της μικροβιακής αντοχής. Η Άγκρη είναι αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή για το θέμα των ε, φαρμακούχων ζωοτροφών με εισηγήτρια την κυρία Αγγιλέρα. Ε, χρειαζόμαστε, και είναι πολύ καλό αυτό το σχέδιο δράση, γιατί θα πρέπει να περιορίσουμε την υπερβολική χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και στα κτηνιατρικά φάρμακα και στα ανθρώπινα ε, γιατί ε, φαίνεται ότι ακριβώς εξαιτία εκτεταμένη χρήση τα, τα αντιβιωτικά γίνονται όλο και λιγότερο αποτελεσματικά για να μην βγούμε και άχρηστα μερικές φορές. Μάλιστα θυμάστε ότι ο Επίτροπος Ανδριουκάητης παρουσίασε το νέο σχέδιο δράσης στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας 13 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Οι Επιτροπές ΕΜΒΗ και ΑΓΡΙ συμφώνησαν να, να παρουσιάσουν έκθεση πρωτοβουλίας με βάση τον, το άρθρο 53 συν και η κυρία Κάντενμπαχ είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Ε, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και είναι και ταυτόχρονα μέρος της Επιτροπής Γεωργίας, κάτι που είναι σημαντικό για να έχουμε συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Ενώ ο κύριος Κάρθη είναι ο συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Άκρη. Και είναι σημαντικό το ότι η κυρία Κάντεμπαχ που είναι η αρμόδια εισηγήτρια της Επιτροπής Εύη είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής Άγκρη. Ε, και σε εμάς είναι ο κύριος Κάρθη, ο υποσυντάκτης της γνωμοδότησης. Ε, ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπω γνωρίζουμε τα μέλη, η αύξηση της ε, μικροβιακής αντίστασης αναγνωρίζεται σαν μία από τις μεγαλύτερες απειλές στην ανθρώπινη υγεία. Μόνο ένα αντιβιωτικό ανακαλύφθηκε τα τελευταία 30 χρόνια και πέρσι το Φεβρουάριο ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας είπε ότι σε μια γενιά χωρί... θα... δεν θα έχουμε... Ε, θα έχουμε προβλήματα, 10 εκατομμύρια κρούσματα προβλημάτων τέτοιων το χρόνο. Οπότε γίνονται όλο πιο σημαντικά τα προβλήματα όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή. Προβλήματα για την κοινωνία, έχει αντίκτυπο και στην ε, οικονομία. Πολλοί γιατροί εξαρτώνται από τα αντιβιωτικά για να αντιμετωπίσουν ασθένειες και μολύνσεις στην ανθρώπινη υγεία και το ίδιο ισχύει και στι εκμεταλλεύσει και οι γεωργοί βασίζονται στα αντιβιωτικά για την υγεία των ζώων, ε, στην κτηνοτροφία και στα, για τα ζώα συνοδεία. Και η χρήση στα ε, κτήματα ήταν τεράστια σημασία για να προστατεύονται τα ζώα και να θεραπεύονται ασθένειε, οι ζωοασθένειε. Οπότε η μικροβιακή αντίσταση ε, χρειάζεται να προσεγγιστεί βλέποντας και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ανθρώπινης υγείας και υγείας των ζώων. Λοιπόν, πρέπει να μειωθεί η χρήση αντιβιωτικών σε εκμεταλλεύσεις και θα πρέπει όμως τελικά να γίνει αυτό χωρίς να επιβάλλουμε μεγάλο εφικοτικό άκθος στους ε, γεωργούς. Είδαμε ότι η αύξηση της γραφειοκρατίας από την πρώτη συζήτηση και του άχθους του διοικητικού στους γεωργούς είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Να αναγνωρίσουμε και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα κόστος, τεράστιο κόστος στην κοινωνία αν χάσουμε την πρόσβαση στα φάρμακα που προστατεύουν την υγεία μας. Τι προσπαθώ να κάνω στη γνωμοδότηση. Να πετύχω σωστή ισορροπία. Όπως προανέφερα, μόνο μια νέα ε, τάξη φαρμάκων ανακαρύφθηκε στα τελευταία 30 χρόνια παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επενδύσει πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε έρευνα για τα φάρμακα από το 1999 σύμφωνα με στοιχεία που έχω πάει από την ε, υπηρεσία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άρα θα πρέπει να ερευνούν και άλλες διεξοδοί άλλε χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία έχουν δημιουργήσει νέες προσεγγίσεις όσον αφορά την κτηνιατρική και θέλουν να μην χρησιμοποιούν μέχρι το 2030 αντιβιωτικά για την υγεία των ζώων. Και θα πρέπει και εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δραστηριοποιηθούμε και να ηγηθούμε και εμεί. Ποιο είναι ο στόχο, βέβαια. Να εξασφαλίσουμε ότι δεν κατηγορούμε απλώ του γεωργού Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την μικροβιακή αντίσταση ξεπερνούν το γεωργικό τομέα, καλύπτεται ε, το θέμα των συνταγών, πωλήσεων, υπερβολική χρήση αντιβιωτικών ψηρά ετών. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Το σχέδιο λοιπόν που έχετε τώρα μπροστά σα ε, καλύπτει νομοθετικέ λύσει ω χρηματοδότηση για του γεωργού, εκπαίδευση, κατάρτιση, σχετικά προγράμματα, αλλαγή όσον αφορά το επιχειρηματικό πνεύμα, αμοιβαία πρότυπα μέσω εμπορικών συμφωνιών, ε, διεθνή συνεργασία κλπ. Λοιπόν, προσβλέπω να ακούσω τι απόψει σα και να συνεργαστώ με του κοιόδη και με άλλα μέλη και ελπίζω τελικά μπορούμε να συνεργαστούμε για να παράγουμε μια καλή συνεισφορά την Επιτροπή και ελπίζω ότι οι συγητή τη ΕΝΒΗ και οι συγητέ τη Επιτροπή ΕΝΒΗ επίση θα λάβουν υπόψη τι απόψει μα. Τώρα, προ ενημέρωση των μελών, προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι 28 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. E, Σας ευχαριστώ πολύ ένα πληρω... οι σκιώδεις εισηγητές Μαγκίνες έχετε το λόγο. Κυρία Μαγκίνες, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή. Νομίζω, ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία για το θέμα αυτό και ότι αποτελεί θέμα ανθρώπινη υγεία. Προφανώς μας απασχολεί πολύ και προφανώ ε, η Επιτροπή Γεωργία έχει γνώμη. Στην παράγραφα την πρώτη, νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίσουμε ότι η χρήση των διαβητικών δεν έχει να κάνει μόνο με τα ζώα, έχει να κάνει και με την ανθρώπινη υγεία. Παράγραφό 2. καλώ ορίζω την έκκληση του κυνηγητή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη για σχέδια δράση. Θα πρέπει οι δράσει αυτέ να λαμβάνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για να πετύχουμε του στόχου που έχουν τέθει. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμό ε, κρατών μελών μεταξύ των Υπουργείων Υγεία και Γεωργία. Στην παράγραφο 3. Για μένα το θέμα αυτό είναι βασικό. Ήδη υπάρχει νομοθεσία που αναφέρεται στα θέματα αυτά, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την, ε, τα φάρμακα. Το 2016 εγκριθήκε η σχετική νομοθεσία. Πάντα μου προκαλεί η νευρικότητα όταν λέμε ότι θέλουμε πιο πολύ νομοθεσία. Όταν υπάρχει η νομοθεσία, είναι απαραίτητο αυτό. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί βασικό μήνυμα στην ε, Επιτροπή Γεωργίας. Ας εφαρμόσουμε αυτά που μόλις έχουμε αποφασίσει και μετά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Στο θέμα της έρευνας, πολύ βασικό, χρειαζόμαστε έρευνα και για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζώα σε θέματα αντιβιωτικών. Υπάρχει το θέμα του κόστου της έρευνα και κατά πόσον οι εταιρείε θα συμμετέχουν. Όλοι πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από ότι η αντιμετώπιση εκ των υστέρων. Και άρα η καλή διαχείριση των ζώων είναι απαραίτητη για να αποθεφεύχονται οι αρρώστιε και οι ασθένειες. Η χρήση των αντιβιωτικών, η παντελής χρήση των, κατάργηση των αντιβιωτικών είναι κάτι ανησυχητικό. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώ Και η παράγραφος 8 είναι παράγραφος κλειδί, θεωρώ κατά πόσον υπάρχει κατάχρηση των αντιβιωτικών. Και πάλι υπάρχει νομοθεσία στη διάθεσή μας. Θα πρέπει τα κρατημέλη απλά να την εφαρμόσουν και να εφαρμόσουν ε, τα συστήματα ελέγχου για να αποφευθεί η κατάχρηση των ε, φαρμάκων. Και τέλος, ε, Θέλουμε μεγαλύτερη συνείδηση για να καταλάβει ο κόσμος τον σύνδεσμο μεταξύ της, σύνδεσης, με της, της υγείας των ζώων και της υγείας των ανθρώπων. βλέπω λοιπόν στις συζητήσεις μας. Σάντος. Σάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Ματ Κάρθη για το σχέδιο γνωμοδότησης και για την παρουσίαση που μας έκανε. Η μικροβιακή εντοχή είναι από τις μείζονες ε, προκλήσεις και παγκόσμια απειλή. Γιατί ο έλεγχος των ασθενειών ε, μερικές φορές αφισβητεί τη χρήση προφυλακτικών αντιβιωτικών. Γι' αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, δυνατότητα χρησιμοποίηση αντιβιωτικών για τις αρρώστιες και όχι προληπτικά και ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία. Είναι τριπλή, τρι, τρεις οι διαστάσεις αυτού του σχεδίου δράσης. Πέραν της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και ε, το περιβάλλον, ε, πρέπει να καταπολεμήσουμε τη μικροβιακή αντοχή. Είναι πλήρης η γνωμοδότηση του κυρίου Ματ Κάρθη και νομίζω ότι με πολύ εύστοχο τρόπο προσεγγίζει τα θέματα του ενίου σχέδιου δράση για την υγεία υπό το πρίσμα της γεωργίας. Επίσης έχουμε τι δεσμεύσει των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης και την ανάγκη ε, θέσπισης κινήτρων προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι. Τα σχέδια δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν ποσοτικοποιημένου ε, καταμετρήσιμου στόχου για να δούμε με βάση τα αποτελέσματα, αν ήταν αποτελεσματικά τα μέτρα που χρησιμοποίησαμε. Επίση, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην διεθνή συνεργασία, είτε μεταξύ των κρατών μελών, είτε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτων χωρών ή περιφερειών. Είναι σημαντικό έτσι να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα, να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση τη μικροβιακή αντοχή. Θα πρέπει να γίνεται συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων και σε θέματα καινοτομία και ανάπτυξης. Θα υποβάλω και κάποιες τροπολογίες και ελπίζω να τις δεχθεί και ο εισηγητής, ο συντάκτης γνωμοδότης και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριος Βάιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Μακάρτη για την καλή πρόταση. Θα ήθελα να αναφέρω από μία ανακοίνωση τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν προαγάγει απαραίτητα τους πράσινους προσανατολισμούς ότι κάθε χρόνο 25.000 ασθενείς χάνουν τη ζωή τους λόγω μικροβιωτικής αντοχής. Στο παγκόσμιο επίπεδο είναι 700.000 αυτά τα άτομα και αυτό μέχρι το 2050 θα μπορούσε να ξεπεράσει ε, το θανατηφόρο παράγοντα και του καρκίνου του ίδιου. Γι' αυτό λοιπόν κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Και να σας πω αυτό πώς σχετίζεται με την γεωργική μας πολιτική. Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι σε βιολογικές ε, αγροκαλλιέργειες 13% ε, των περιπτώσεων έχουν να κάνουν με μικροβιατική αντοχή ενώ ουσιαστικά στις ε, σημαντικές καλλιέργειες είναι 50% αυτό το ποσοστό. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εξηγήσουμε και στον κύριο Ακνιού τι γίνεται στη βιομηχανική καλλιέργεια. 70% όλων των επιχειρήσεων έχουν τέτοια α, πολύ ανθεκτικά μικρόβια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόβλημα υπάρχει και αυτό μπορεί να μας υποδείξει τι επιχειρήσεις θέλουμε να υποστηρίξουμε με τις ε, ευρωπαϊκούς πόρους και πώς μπορούμε να προαγάγουμε την ευρωπαϊκή υγεία. Αγγουλέρα. Κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Κάντεμπαχ που παρόλο που θα ήθελε πολύ να παρακολουθήσει τη συζήτηση έπρεπε οπωσδήποτε να φύγει. Ε, ευχαριστή κυρία Κάντεμπαχ τον κύριο Κάρθη για την γνωμοδότησή του που είναι πολύ καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση στην Επιτροπή και θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία της γνωμοδότησης του κυρίου Ματ Κάρθη. Ε, συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνες ε, σε ό,τι αφορά την απέτηση για νομοθετικές λύσεις. Εγώ έχω μεγάλες προσδοκίες από τα εθνικά σχέδια δράσης, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό και κάποια, κάποιο monitoring μετά, κάποια παρακολούθηση και ήδη έχει ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία για τη σχετική πρόταση σε ό,τι αφορά τις φαρμακούχε ζωοτροφές και τα κτηνιατρικά φάρμακα. Εμείς είμαστε πολύ πιο γρήγοροι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο καθυστέρησε κάπως. Τώρα ξεκινούν οι τριμεροί διάλογοι για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Οπότε θα έχουμε και νομοθετικές διατάξεις που θα διέπουν τη χορήγηση αυτών των ουσιών και τον έλεγχο για να μειώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία. Και ευελπιστώ ότι ως ονόπο θα έχουμε δύο κανονισμούς. Έναν για τις φαρμακούχες ζωτροφέ και ένα για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Και Ελπίζω να έχουμε και άλλο ένα παρόμοιο και τρίτο νομοθέτημα, ώστε να έχουμε ένα επαρκές φάσμα νομοθετικό για να καλύψουμε τη μικροβιακή αντοχή. Γιατί ε, δεν κρίνω σκόπιμο να ζητήσουμε νέε νομοθετικέ προτάσει. Ήδη υπάρχουν αρ, και επίσης έχουμε και τα εθνικά σχέδια δράσης. Και σημαντικό είναι να επενδύσουμε στην έρευνα στην επιστημονική έρευνα, γιατί χωρίς επιστημονική έρευνα δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Πιστεύω ότι από νομοθετική άποψη ό,τι έχουμε είναι καλό, θα πρέπει να το προωθήσουμε και επίσης ε, ε, η ανάπτυξη πιο αηφόρων συστημάτων παραγωγής. Αηφόρων μεν, ανταγωνιστικό δε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητα, να δώσουμε έμφαση στην αηφορία, αλλά όχι ερήμην της ανταγωνιστικότητας. Γιατί αν οι δεν έχουν κερδοφόρο δραστηριότητα θα εγκαταλείψουν την κτηνοτροφία. Οπότε θέλουμε αηφορία, μην ξεχνούμε και την ανταγωνιστικότητα. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντική η ανταγωνιστικότητα με την αηφορία. Επίσης δεν συμφωνώ και πολύ με τον ορισμό στο σημείο 8. Πιστεύω θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή νοοτροπίας και ε, να χρησιμοποιούμε γενικώ λιγότερα αντιβιωτικά και στα ε, φάρμακα για, τους, ε, για την ανθρώπινη χρήση αλλά και στα κτηνιατρικά φάρμακα. Και πραγματικά δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούνται εκτεταμένο στα κτηνιατρικά φάρμακα ή φαρμακούχες μόνο για την προσπόρηση κέρδους. Αυτό είναι άδικο, όπως το λέει ο εισηγητής στο σημείο 8. θα πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία και να χρησιμοποιούμε λιγότερα αντιβιωτικά και οι άνθρωποι και φυσικά και οι κτηνοτρόφοι για τα ζώα που εκτρέφουν. Αλλά δεν γίνεται συστηματική χρήση τους στη μαζική παραγωγή. Και συμφωνώ να δώσουμε έμφαση στην αηφορία, αλλά ταυτόχρονα και στην ανταγωνιστικότητα, για να μην εξαφανιστούν οι κτηνοτρόφοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Σάγνιου. Ευχαριστώ. Πραγματικά σημαντικό, σημαντικό θέμα. Όλοι ξέρουμε κόσμο που δεν θα ζούσε σήμερα αν δεν υπήρχαν τα αντιβιωτικά και αν γίνουν τα μικρόβια ανθεκτικά, θα πεθάνει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό να το συζητάμε. Ποια είναι η απόψή μου. Εγώ ασχολούμαι με τα πουλερικά και την παραγωγή αυγών. Μιλάμε για τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτή είναι σωστή προσέγγιση πιο κοντά στη φύση και αυτό είναι καλό, λένε όλοι. Να είναι ένα πρόβλημα που έχουμε εμείς. Ανακαλύψαμε ότι μολυνόταν το σύστημα ποσίμου υδάτων, ε, δημιουργούσε προβλήματα και δύσκολο να εκναρετήσουμε πώς μολυνόταν το νερό με ακαθαρσίες και μπήκε σωλήνες ποσίμου. Τέλος πάντων το λύσαμε. Τι ανακαλύψαμε. Αφήναμε το πρωί να βγουν τα πουλιά και πήγαιναν στην λιμνούλα την πιο κοντινή που ήταν μολυσμένη. Αυτό κάνουν. Πάνε και κολλάνε, παθαίνουν διάφορες ασθένειες από αυτά τα βρώμικα νερά. και μετά από τέσσερις μήνες βροχής ε, και λοιπά, πάνε εκεί το χειμώνα. Εμείς λέμε στον κλινίατρο να κρατήσουμε τα πουλιά μέχρι το μεσημέρι μέσα, να φάνε, να πιούνε το νερό τους μέσα το καθαρό νερό και μετά να τα αφήσουμε να βγουν. Όμω αυτό είναι κατά των κανόνων περί κοτόπουλων, κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής. Να προβλήματα πραγματικά αυτά. Έχουμε ένα πρόβλημα. Πάμε στον κτηνίατρο με ένα νεκρό πουλί. Ε, μας προτείνουν κάποιο αντιβιωτικό, το βάζουμε στο νερό και ξαφνικά μέσα σε δύο εβδομάδες αυξάνεται η παραγωγή αυγών και μειώνεται η θνησιμότητα. Αν δεν μπορούσα να το κάνω εγώ αυτό, δεν θα μπορούσα να δουλέψω καθόλου. 150.000 λίρες το χρόνο μου κοστίζει να αγοράζω τα πουλερικά μου και να αρρωστήσουν τα πουλερικά γιατί δεν μπορούσα να τα θεραπεύσω με αντιβιωτικά ε, με κάνει να, ε, να φρύτω, δεν μπορώ να αντέξω καν τη σκέψη. Τι μπορεί να γίνει. Χαίρομαι ο κύριος Κάτες ανεφέρθηκε στο, στο θέμα. Αν ένας νόμος λέει, κύριε Άγνιου, ου χρησιμοποιήσει αντιβιωτικά είμαι εκτός συστήματος εγώ. Αν υπάρξει και κάποιο καρότο πέρα από τη ράβδο. Αντί να μου λέει αυτό, το ου, οι πληρωμέ του πυλώνα 1 πάνε στο φίλο σα στην Ιρλανδία, πώ τον λένε. Τέλο πάντων, υπάρχει ένα ταμείο, ούτω ώστε κάποιο πρέπει να αποφασίσει. Θα χρησιμοποιήσω αντιβιωτικά ή θα σκοτώσω τα πουλερικά. Δεν μπορεί να αφήσει κανεί την κατάσταση ω έχει είναι θέματα ευζοίας των ζώων και λοιπά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μπορούμε να αφήσουμε τα πουλερικά να στενούν. Οπότε θα θανατώνεις τα πουλερικά και παίρνει κάποια πληρωμή. Τέλο πάντων, γρήγορο, συγγνώμη Πρόεδρε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορο. Χρειαζόμαστε υποστήριξη από τι υπεραγορέ, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε ε, το δρόμο τη μη χρήση αντιβιωτικών. Πρέπει να υποστηρίξουν τι εκμεταλλεύσει που το κάνουν αυτό. Και τι γίνεται τώρα με την αναπαραγωγή. Υπάρχουν ε, θέματα αντοχής και αντίσταση μια ασθένεια. Υπάρχουν άγρια πτηνά που είναι αρκετά ανθεκτικά σε προβλήματα για τα οποία εμεί χρειαζόμαστε αντιβιωτικά. Έχουμε τεχνολογία, μπορούμε να πάρουμε τα γονίδια από τα, τα ελεύθερα πουλιά, να τα βάλουμε στα κοτόπουλα και θα εμβολιάζονται και θα αντέχουν σε αυτές τις ασθένειες και θα θεραπεύονται. Ας το σκεφτούμε και αυτό. ναι, ε, ναι αλλά το το κατόφλι ανοχή στην παράβαση του χρόνου αγόρευσης είναι άλλο θέμα. Ο κύριος ε, Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συζήτησα αυτό το θέμα με χειροτρόφους και πτυνοτρόφους και τους ρώτησα πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα της ε, κατανάλωσης ε, κτηνιατρικών φαρμάκων. Ε, η απάντησή τους ήταν ότι χρησιμοποιούν ελάχιστα, σχεδόν καθόλου φάρμακα στην κτηνοτροφία και κατάφεραν να ελέγξουν τη χρήση αντιβιωτικών εξασφαλίζοντας ε, καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων ε, στις μονάδες τους. Και σας διαβεβαιώ ότι 80% των κτηνοτρόφων 80% μάλλον των αγροτών ε, ζούσαν σε χειρότερες συνθήκες διαβίωσης από ό,τι τα ζώα στις ε, κτηνοτροφικές μονάδες και γι' αυτό δεν χρειάζονταν ε, αντιβιωτικά. Νομίζω ότι οι καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων και κίνητρα για την ευημερία των ζώων θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών ή αντιμικροβιακών ουσιών. Άλλοι τώρα κτηνοτρόφοι που έχουν αγελάδες, βοηθοί άλλα ζώα που προτιμούν ε, ε, αντί να χρησιμοποιούν φαρμακευτική αγωγή να σκοτώνουν τα ζώα γιατί το, ε, το τίμημα της φαρμακευτικής αγωγής είναι πολύ ψηλό. Τι να πω. Πιστεύω ότι δίνοντας έμφαση στην ευημερία και στις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων θα περιορίσουμε τη χρήση αντιβιωτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αλλά παρακαλώ να είστε πιο λακωνικοί. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω και είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, αυτό το θέμα είναι τεράστια έκταση και η χρήση αντιβιωτικών, η ε, εφεύρεση των αντιβιωτικών ήταν μία από τις ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τη ανθρωπότητα. και είχε τεράστια διαγετήματα για την ανθρωπότητα. Το βλέπουμε και στους εαυτούς μας και στα σχολεία. Μου το λένε όλοι οι δάσκαλοι, όλων μου των παιδιών, ότι ποτέ δεν έχουν δει τόσα πολλά παιδιά να λείπουν από το σχολείο και δεκάδες, ε, μάλλον δόσεις ε, επιδόσεων ε, φαρμάκων δεν έχουν αποτέλεσμα και αυτό μας δείχνει σε τι βαθμό επικεντρινότητας ήδη έχουμε βρεθεί. Στην τελική ανάλυση ο αγρότης δεν θέλει να βλάψει προφανώς κανένα άνθρωπο και την υγεία του. Θέλουν να παράγουν καθαρή τροφή, καθαρά τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Και εδώ λοιπόν το αντίπαλο δέος είναι ότι οι αγρότες πρέπει να βγάζουν τα προς το ζήντ και προφανώς έχουν κόστος. Αν ακολουθήσουμε αυτή τη λογική και αυτή τη λογική θα πρέπει να ακολουθήσουμε για την άμα, υπερβολική χρήση των αντιβιωτικών, αυτό θα έχει πολύ προφανώς ένα κόστος πολλά θα είναι τα μειονεκτήματα του Brexit. Ο κύριος Νικόλσον και ο κύριος Αγνιού μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες και θα μας λείψουν. Είναι πάρα πολύ ενημερωτικά αυτά που μας λέτε. Είναι γεγονός ότι μπορεί κανείς να αγοράσει βιολογικά αυγά που δεν έχουν αντιβιωτικά, αλλά πολύ απλά κοστίζουν παραπάνω. Και ξέρω ότι λίγο πολύ όλοι οι γονείς στη χώρα μου και στην περιοχή μου αγοράζουν αυτά τα αυγά. Μάλλον θα τα αγόραζαν σίγουρα εάν δεν κόστιζαν πιο πολλά λεφτά. Άρα η πρόληψη είναι καλύτερη παρά η θεραπεία, προφανώς. Αλλά η πρόληψη στην περίπτωση αυτή θα κοστίσει. Αν είναι λοιπόν να επιμείνουμε στην πρόληψη, θα χρειαστούμε χρήματα. Δεν μπορεί να είναι αυτό ει βάρος των όσων παράγουν τα τρόφιμα. Και αυτό θα κοστίσει με τη σειρά του χρήματα. Ποιο θα τα πληρώσει αυτά τα χρήματα, ο κ. Χόισλινγκ. Ευχαριστώ για την έκθεση. Είμαι σκιώτη. Για τα ακτινητικά σκευάσματα. Και είμαστε στο δεύτερο τρομερή διάλογο. Νομίζω από πλευρά του Κοινοβουλίου έχουμε καταρτήσει αφήσεις κανόνες για τα αντιβιωτικά και την αντιβιωτική κατάχρηση που συνδέεται και με την εκτροφή των ζώων που δεν είναι ιδανική. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε, το είπε και ο συνάδελφος, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε και με επικριτικό τρόπο τη χρήση αντιβιωτικών Το είπε και ο συνάδελφος ότι έφερε και θέμα ανταγωνισμού. Θα πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι δεν θα ωφελήσουμε την ε, συνολική κοινωνία αν ε, βάλουμε την ανταγωνιστικότητα, το φτηνό κρέας πάνω από το συμφέρον των μελλοντικών γενιών, την επιβίωσή τους. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει. Πρέπει να παράγουμε κρέας, μάλιστα. Αλλά δεν μπορούμε να μελήσουμε θέματα επιβίωσης. Και σε άλλο βαθμό μπορούμε να επιμείνουμε σε ό,τι αφορά τη μείωση. Το θέμα της ε, μεταφυλακτικής σε ό,τι αφορά τα, τη μικροβιακή αντοχή. Αυτό τι σημαίνει ότι ε, ασθενεί ένα τμήμα των ζώων και προφυλακτικά δίνουμε διευθυντικά στα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και πάντα με εκνευρίζει γιατί τελικά το φρένα το πατούν τα κράτη-μέλη για να προστατεύσουν προ... τα συμπέροντα του κλάδου. Εμείς ως κοινοβούλιο θα πρέπει να χαράξουμε το δρόμο του μέλλοντος και πού θα πρέπει να επιμείνουμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι είμαστε οι μοναδικοί εδώ στην Ευρώπη που θέλουμε να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πολύ απλά μας έχουν παραδείσει. Ο κύριος Χόιμπος. Η κυρία Χόιμπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη ακούσαμε. Και ο κύριος είπε, νομίζω, το πιο ουσιώδες. Είπε ότι πολλοί κόσμος δεν θα ζούσε αν δεν υπήρχαν τα αντιβιωτικά. Δεν θα ζούσε αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα αυτό. Όταν μιλάμε για πολυανθεκτικά βακτήρια, αυτό τι σημαίνει ότι δεν έχουν επίδραση τα αντιβιωτικά μας και εδώ τα εφεδρικά αντιβιωτικά έχουν ιδιαίτερο ρόλο. Η προστασία του ανθρώπου θα πρέπει να υπερισχύει της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας του ζώου. Όταν έχουμε και επιτρέπουμε εφεδρικά αντιβιωτικά λοιπόν, σε κάποια χρόνια πολύ απλά δεν θα χρειάζεται να μιλάμε τα εφεδρικά, να μιλάμε για τα εφεδρικά αντιβιωτικά, δεν θα υπάρχουν. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ναι, όντως αυτή την άποψη θα πρέπει να την διαδώσουμε και να τη λάβουν υπόψη και οι πολιτικοί θύνοντες. Και οι πολιτικοί θύνοντες θα πρέπει να νιώσουν τη σοβαρότητα του προβλήματος. Ο κύριος Ντές. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Το θέμα αυτό προφανώς θα πρέπει να το κοιτάξουμε με μεγάλη προσοχή, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θα πρέπει να αντιπιστώσουμε και ποια είναι τα περιστατικά και τα γεγονότα. Σε ό,τι αφορά την εκτροφή των ζώων έχουμε πολύ αυστηρές προδιαγραφές στη Γερμανία και όντως ισχύει η χρήση των αντιβιωτικών από το 2011 μέχρι το 2015 μειώθηκε κατά το ίμιση και πλέον. Η Γεωργία λοιπόν θεωρώ ότι συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Στη Γερμανία έχουμε μία υπουργό έχουν το, με το Ινστιτούτο για την Αξιτήμηση των ε, Κινδύνων και το 2012 τότε ήδη διαπίστωσαν σε έρευνες ότι τα πολυεθνικά βακτήρια στα νοσοκομεία έχουν σε 5% αιτία στη γεωργική καλλιέργεια και στις εκτροφές και μόνο κατά, μόνο κατά 5% και 95% από, άλλους, ε, από άλλες Ύστερα, σε ό,τι αφορά τη χρήση των αντιβιωτικών, ε, η θεραπεία έχει περιοριστεί εκτοτε από 5 σε μία ημέρα. Εδώ λοιπόν διαπιστώνουμε ε, θετικέ αλλαγές. Επίσης, τι γαλακτοκομικές επιχειρήσεις. Κάνουμε αντικμεταλλευτικού ελέγχους κάθε μέρα. Κάθε μέρα, επαναλαμβάνω. Η προστασία λοιπόν του ανθρώπου είναι απόλυτα εκγυημένη. Άρα εγώ τι να σας πω, δεν πιστεύω και πραγματικά ανίσταμε όταν λέμε ότι η Γεωργία ευθύνεται για όλα. Από την Γενική Διεύθυνση Υγείας, ο κύριος Ρίκτε δεν έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά χαιρετίζει την ιδιαίτερη προσοχή που δίδεται στο ζήτημα της μικροβιακής αντοχής γιατί όπως ξέρετε η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής είναι προτεραιότητα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως φαίνεται και στο σχέδιο δράσης που εθέτησε στα μέσα του περασμένου έτους. Είναι σημαντικό λοιπόν να εγκύψει το θέμα αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι κοινή μας ευθύνη και θα πρέπει να διέπει όλες μας τις ε, δράσεις ε, να έχουν στόχο την, ε, τον περιορισμό της χρήσης των αντιβιωτικών. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Άγκρη, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Ήδη άρχισαν οι τριμερείς διάλογοι σε ό,τι αφορά τις προτάσεις κανονισμών για τις φαρμακούχες ζωοτροφές και τα κτηνιατρικά φάρμακα. Χάρη στις συζητήσεις αυτές ε, θα ε, αντιμετωπίσουμε και πολλά θέματα που επισημαίνεται στο σχέδιο γνωμοδότηση. Για παράδειγμα, την ε, απαγόρευση της προληπτικής χρήσης αντιβιωτικών ή τον περιορισμό ε, της προφύλαξης ή μεταφύλαξης που ε, προέκυψε και στη συζήτηση. Επίσης, θα γίνουν συζητήσεις για τον περιορισμό ε, της διαφήμισης ή της ε, διάθεσης των ε, φαρμάκων. Όλα αυτά τα θέματα που θα συζητηθούν στις τριμερείς διαλόγους πιστεύω ότι θα καλύψουν και τις δικές σας ανησυχίες όπως προκύπτουν από την γνωμοδότηση. Ό,τι αφορά την υποστήριξη που θα δώσουμε στους αγρότες σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ΚΑΠ και το, της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης υπάρχουν διάφορα ε, μέσα στήριξης όπως ε, ε, ενίσχυση των επενδύσεων, στήριξη στις επενδύσεις σε περίπτωση που οι κτηνοτρόφοι θέλουν να βελτιώσουν την ασφάλεια στην κτηνιατρική μονάδα τους ή να βελτιώσουν ε, τις συνθήκες των ζώων ή να περιορίσουν τη χρήση αγωγής ή αντιβιωτικών φαρμάκων τα ίδια μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα πλαίσια της κατάρτισης ή της ευαισθητοποίησης. Για να βοηθήσουμε λοιπόν τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους ε, να χρησιμοποιήσουν τις συμβουλές που προσφέρουν τα κράτη-μέλη στα, πλαίσια κάποιων προγραμμάτων παροχής συμβουλών σε επίπεδο ε, εκμετάλλευσης ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση αλλά και η κατάρτιση σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Και τέλος, το θέμα ε, του παγκοσμίου επίπεδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προασπίζει τη θέση της και τη θέση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και διεθνώς. Ε, θέλουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο να ε, με το ενδιαφέρον και την προσοχή στα θέματα της μικροβιακής αντοχής προκειμένου να έχουμε κάποιες ε, διεθνείς πρωτοβουλίες όπως είναι ο κώδικας ε, στο Διεθνή Οργανισμό και όταν έχουμε εμπορικές διαπραγματεύσεις με εταίρους, εμπορικούς εταίρους και εκεί επισημαίνουμε τη σοβαρότητα που έχει η μικροβιακή αντοχή και προσπαθούμε να τους πείσουμε για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της χρήσης αντιβιωτικών προληπτικά. Οπότε και στις εμπορικές μας διαπραγματεύσεις υιοθετούμε παρόμοια στάση. Αυτά λίγο πολύ είχα να πω. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για τις προτάσεις και θα συνεχίσουμε τον κοινό μας αγώνα κατά Τη μικροβιακή αντοχής, τη αυξανόμενη δυστυχώς αντοχής των μικροβίων στα φάρμακα. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρθη τώρα, ο συντάκτη γνωμοδότη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ του συναδέλφου και τα σχόλια. Κουβάντιζα με τον παθολόγο μου σε κάποια φάση εδώ και χρόνια. Μου έλεγε, Όλοι θέλουν οι άλλοι να μην χρησιμοποιούν τα αντιβιωτικά. Όταν αρρωστήσουν αυτοί θέλουν τα αντιβιωτικά. Άρα έτσι αντιλαμβανόμεθα το πρόβλημα. Ποια είναι η αλήθεια. Πρέπει να μειώσουμε τη χρήση αντιβιωτικών. Η γνωμοδότηση δεν ζητά απαγόρευση χρήσεως αντιβιωτικών. αναγνωρίζει τη σημασία των αντιβιωτικών, ότι παίζουν σημαντικό ρόλο για τα ζώα, για την ευημερία των ζώων. Οι κτηνοτρόφοι σε κάποιο επίπεδο θα εξακολουθούν να δίνουν αντιβιωτικό δεδομένο. Πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι μειώνεται το επίπεδο αυτό και ότι χρήση τους γίνεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο. Κατανοώ τα σχόλια και τις απόψεις που εκφράστηκαν σχετικά με την παράγραφο 3 Ποια είναι η αλήθεια. Ότι οι φαρμακοζώτροφες είναι ένα θέμα για το οποίο είμαι και εκεί συντάχτης κειμένου. Συνεχίζονται οι εργασίες, είμαστε σε τριμερή διάλογο. Στόχος της παραγράφου 3 είναι να καθορίζουμε σαφέστατα ότι είναι πρόθυμη η Επιτροπή να εξασφαλίζει την εφαρμογή βελτίστων πρακτικών. και να λαμβάνεται υπόψη η εντολή μας και το τομέα μας. Στα πλαίσια της γενικής προσεγγίσεως για την υγεία. Δεν θέλουμε να κλείσουμε καμία εκμετάλλευση του κυρίου Άγνιου του κανενός άλλου. Πράγματι. Χρειάζεται προσέγγιση καρότου και ραβδιού. Πρέπει να στηρίξουμε τους γεωργούς και τον ευρύτερο τομέα για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων, αλλά πρέπει να προστατεύουμε και τους ανθρώπους και τα ζώα από την υπερβολική χρήση αντιβιωτικών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα επίπεδα της μικροβιακής αντοχής θα μειωθούν. Θα συνεργαστώ με τους κοιόδης και με όσους άλλους υποβάλλουν τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να εξασφαλίσω ότι θα έχουμε γνωμοδότηση της Επιτροπής που θα είναι ευρεία με πολιτική υποστήριξη στο βαθμό του δυνατού στην Επιτροπή, ούτω ώστε με ισχυρά επιχειρήματα να πάμε και να συμπληρωθούν συστάσεις νομοδοτήσεως στην έκθεση της ΕΜΒΙΑ όπως αναφέρθηκε από πολλούς ομιλητές, τους οποίους ευχαριστώ, όπως είπαν λέγω, είναι τεράστιο θέμα, πιθανότατα καθοριστικό θέμα της εποχής μας. Έχουμε όλοι ρόλο να παίξουμε και η κοινότητα των Γεωργών και αυτή η Επιτροπή μπορεί να παίξει παραγωγικό ρόλο κατευθύνοντας ε, τις σωστές δράσεις εκεί που απαιτούνται. Ευχαριστώ. Θέλουμε και περισσότερη γνώση και περισσότερες πληροφορίες και περισσότερη συνειδητοποίηση και στο επίπεδο των κτηνοτρόφων αλλά και πιο πέρα. Γιατί οι κτηνοτρόφοι είναι παραγωγή τροφίμων. Παραγωγή τροφίμων σημαίνει διατροφή. Διατροφή σημαίνει υγεία. Είναι πολύ διάστατο λοιπόν το φαινόμενο και συμφωνούμε με τον εισηγητή Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου στη 1 το μεσημέρι έχετε διορία για την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστούμε τον συντάκτη γνωμοδότη, ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχαριστούμε τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση και να περάσουμε στην έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Τις λάβατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και ε, γράφος. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις τις εγκρίνουμε και ολοκληρώνουμε εδώ μια πολύ γεμάτη και πολύ άσχολη εβδομάδα. Είχαμε πολλά θέματα και εκείνη η γεωρική πολιτική και το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, τον οικολογικό προσανατολισμό, την υγεία, πλούσιο πρόγραμμα είχαμε αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο. Μην, ξεχά, μην ξεχνάτε να στέλνετε τις ερωτήσεις προς τον κύριο Ντόφμα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.